Okay. Uh, welcome back. We will now continue the... Καλώς ήρθατε και πάλι. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα ξεκινήσουμε τώρα. Κοινή ακρόαση της Επιτροπής Γυναικών και της Επιτροπής ε, ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Χαίρομαι που έχω εδώ στο πλευρό μου τον κύριο Αγγιλάρ και που θα πραγματοποιήσουμε μαζί ε, την σημερινή ακρόαση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι θέμα που αφορά και τις δύο επιτροπές. Χαίρομαι λοιπόν πολύ για αυτό. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Αγγιλάρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκούσταυσον. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμπροεδρεύω εδώ σε αυτήν την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελίμπε και της Επιτροπής Γυναικών. Σας καλωσορίζω λοιπόν σε αυτήν την κοινή ακρόαση για τις ε, εθνικές στρατηγικές ένταξεις των Ρωμά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτών. Είναι ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας και για τις δύο αυτές επιτροπές του Κοινοβουλίου και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ' αυτό, διότι εκφράζει μία μόνιμη δέσμευση προς τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Η ένταξη ούσα ένα από αυτά ισότητα και ισονομία και κατάργηση των φραγμών στο δρόμο της ισότητας. Αυτό είναι ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα που θα μας απασχολεί για πολύ καιρό. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ορισμένους ε, εξειδικευμένους καλεσμένους που θα μας παρουσιάσουν την ε, αναλυτική πρόοδο και τις στρατηγικές ένταξεις των ε, πληθυσμών Ρωμά, τις εθνικές στρατηγικές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι μία απάντηση σε μία κατάσταση που για πολύ καιρό αγνοούσαμε. Οι διακρίσεις κατά των ε, Ρωμά δεν ήταν πάντα κάτι το αρκετά ορατό στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή εκπληρώνουμε τις ε, υποχρεώσεις που έχουμε για να το κάνουμε το ζήτημα αυτό ορατό και να το καταπολεμήσουμε. Πέρυσι το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμά του ζήτησε ξεκάθαρες, έκανε ξεκάθαρες συστάσεις στα κράτη-μέλη και ζήτησε την ε, εξάλληψη των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά, των εξώσεων, των διακρίσεων και ζήτησε από τα κράτη-μέλη να δώσουν μια κατάλληλη λύση για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των Ρωμά με ξεκάθαρες προπτάσεις. Αξιολόγηση και παρακολούθηση των διάφορων project για τις κοινότητες ε, Ρωμά και χρησιμοποίηση όλων των δυνατών ευρωπαϊκών πόρων. Τέλος, ένα χρόνο μετά από την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών θεωρούμε πως έχει έρθει η ώρα να αξιολογήσουμε και τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού αυτού πλαισίου και της προόδου που έχει επιτευχθεί σε καθένα από τα κράτη-μέλη και να δούμε τι άλλο χρειάζεται να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλιστεί το, ο απόλυτο σεβασμός όλων των ε, δικαιωμάτων των Ρωμά σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ε, εκ των προτέρων. Ευχαριστούμε πολύ τους ε, καλεσμένους που θα ακούσουμε σήμερα. Και αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ακούσουμε μία παρουσίαση από την κυρία Γιαρόκα, εισηγήτρια της Επιτροπής Γυναικών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω όλους σας και σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο πολύ εδώ. Νομίζω ότι η συνάντηση είναι πολύ σημαντική γιατί θα ακούσουμε μαρτυρίες από Ρωμά και μη Ρωμά για το τι γίνεται στην Ευρώπη στην εφαρμογή και υλοποίηση της στρατηγικής για τους Ρωμά. Αύριο θα πάμε σε μια αποστολή στην Ουγγαρία και την Κροατία για να δούμε πώς είναι η κατάσταση επιτόπου. Δεν πρόκειται για επίσημη αποστολή του Κοινοβουλίου. Δεν έχει γίνει επίσημη αποστολή του Κοινοβουλίου ποτέ σε Ρωμά. Και θα πάμε να δούμε την πραγματικότητα εκεί. Θα ακούσουμε από τους ανθρώπους, από, την, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, τι κάνει ο κάθε φορέας για να καταλάβουμε την κατάσταση καλύτερα καλέσαμε και εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των νοικιόπου που δραστηριοποιούνται στον χώρο για να μας δώσουν μια εικόνα των τελευταίων ευρημάτων βάση των εθνικών προγραμμάτων δράσης, της πρόοδου που είδαμε επί τόπου και του τρόπου αξιολόγησης των μέτρων αυτών από τους ε, ε, εμπλεκόμενους και με χαρά ε, δεχθήκαμε διάφορες ομάδες επισκεπτών από διάφορες χώρες της Ένωσης και την Ουγγαρία που νομίζω ότι θα μπορέσουν να δώσουν πραγματική ενημέρωση για να συμπληρώσουν τη συζήτηση στα θέματα που συζητούμε. Το σημαντικότερο στοιχείο της έκθεσης είναι ότι διερευνά τα προβλήματα. Ξεκινά ως μια κριτική δράση, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει συστάσεις και έχουμε λόγο στα έγγραφα της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θέλουμε τώρα να προχωρήσουμε παραπέρα. Να έχουμε σαφείς δείκτες και ένα πλαίσιο ελέγχου που θα στηρίζεται στους δείκτες αυτούς και που θα καταστήσουν το πρόγραμμα, τα προγράμματα χρήσιμο, χρήσιμα και όχι απλά κουβέντες. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στα απτά αποτελέσματα. Εγώ ως Ουγγαρέζα έχω εμπειρία από πρώτο χέρι για την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας συμφώνησε και με τους Ρωμά και με τις ΜΚΟ να υπάρχουν ποσοτικοποιημένα μέτρα. Ποσοτικοποιημένα μέτρα. Στα κράτη-μέλη η στρατηγική λύπη. Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε μεγάλα προγράμματα εκπαίδευσης, μεταρρύθμισης εκπαίδευσης ή απασχόλησης δεν ενσωματώνεται η διάσταση της στρατηγικής κατά της φτώχειας. Δεν βλέπουμε τα κράτη-μέλη να έχουν οικονομικά προγράμματα που θα προσανατολίζονται στα θέματα των Ρωμά. Κατέστη σαφές επίσης, και μπορεί να το πει η Επιτροπή, ότι η εμπλοκή ΜΚΟ και πολιτών είναι εξαιρετικά αδύναμη. Ο κύριος στόχος δεν επιτυγχάνεται. Οι ΜΚΟ δεν αντιπροσωπεύουν στόχους που θέλουν οι πολίτες. Ο διάλογος δύσκολα υλοποιείται, δεν υπάρχουν βήματα διαλόγου συχνά. Τώρα είναι μια περίπτωση. Απλά να σας πω εν γέννη ότι οι ΜΚΟ δεν εμπλέκονται σοβαρά στο θέμα. Επίσης έχουμε ένα χάρτη κρίσης, μια περίπτωση κρίση στην, μια περίοδο κρίση στην Ευρώπη. Υπάρχουν κέντρα αντιμετώπιση κρίση στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες όπου υπάρχει εγκαιτοποίηση, στην Πορτογαλία για παράδειγμα, χωρίς να υπάρχουν μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπίσουν αυτά τα μαζικά προβλήματα άτομα που ζουν στην φτώχεια, στις, ε, στους καταβλισμούς αυτούς, χωρίς να βλέπουμε συντονισμένη δράση. Και το τελευταίο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι κατά την άποψή μου, τουλάχιστον όσο βλέπω, το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε πέρσι δεν δίνει σωστές απαντήσεις. Δεν καλύπτει επαρκώς. Τα εθνικά σημεία αναφοράς πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα, να υπάρχει μια πραγματική συζήτηση και να, εκτεθούν, να εκτίθενται οι κακές πρακτικές. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα που θα πρέπει ωστόσο να μπορούν να δώσουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Τελειώνω εδώ. Ευχαριστώ κυρία Γιάροκα. Να ακούσουμε τη συνάδελφό μας ε, κυρία Κίνκα Δεν ε, θέλω να μακρηγορήσω διότι σήμερα κυρίως θέλουμε να ακούσουμε τις εμπειρίες άλλων. Αλλά θα ήθελα να πω ότι όπως το βλέπω το πιο σημαντικό επίτευγμα είναι ότι έχουμε σε εθνικό επίπεδο αυτές τις στρατηγικές ένταξεις των Ρωμά. Δεν ε, βλέπουμε όμως πάντα τη χρηματοδότηση ούτε την πολιτική βούληση ε, και γι' αυτό έχω καλέσει σήμερα εμπειρογνώμονες που θα μας πούνε σε τι βαθμό υπάρχει τέτοια πολιτική βούληση ενδιαφέρον για μένα είναι ότι από τη μία έχουμε αυτά τα έγγραφα, ελπίζω να μην είναι απλά κενά έγγραφα, από την άλλη έχουμε ε, πολιτικές αποφάσεις ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Μερικές φορές βλέπουμε οι πραγματικές πολιτικές αποφάσεις και οι στρατηγικές ένταξεις των Ρωμά ε, να μην έχουν ε, καμία σχέση μεταξύ τους. Στο κράτος μέλος που γνωρίζω καλύτερα, την Ουγγαρία, Βλέπουμε ότι νομιμοποιείται όλο και περισσότερο αγώνας κατά των διακρίσεων. Ε, Βλέπουμε ότι αυξάνεται το επίπεδο της εκπαίδευσης, κάτι μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη θέση απασχόλησης αργότερα. Μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση όσον αφορά την φτώχεια. Επίσης έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι θα πρέπει οι ευρωπαϊκοί πόροι να ε, βοηθήσουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε αναμορφωτήρια νέων ε, αντί να ε, ε, αντί για καλύτερη εκπαίδευση που θα οδηγήσει σε καλύτερη θέση απασχόλησης στο μέλλον σε επικοινωνιακό επίπεδο βλέπουμε λοιπόν μια αρκετά ρόδινη εικόνα, ε, σε κοινωνικό επίπεδο βλέπουμε το αντίθετο μάλλον. Ε, θα ήθελα λοιπόν πολύ να ακούσω περισσότερα από τους εμπειρογνώμονές μας ε, που θα μας μιλήσουν για την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια σκιώδη έκθεση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τις δύο πλευρές, δηλαδή τις κυβερνητικές εκθέσεις, την έκθεση της Κομισιόν και τις εκθέσεις των ΜΚΟ συχνά ε, έχει κανείς την εντύπωση ότι μιλούν για τελείως διαφορετικά μέρη του κόσμου. Μία σύντομη παρατήρηση για την Επιτροπή της ΕΦΕΡΑ. Ε, είναι σαφές ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και σημαντική έλλειψη ε, στοιχείων, δεδομένων που είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλοι από εμά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιες καλές πρακτικές και κάποιες κακές πρακτικές. Ποια είναι όμως η πραγματική κατάσταση. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που να προσανατολίζεται περισσότερο στα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα και πιστεύω ότι και τα κράτη-μέλη έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να πιέσουν δηλαδή τα κράτη-μέλη. Είμαι βέβαιη ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουμε οργανώσεις των Ρωμά, διότι αλλιώς δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο που πρέπει. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο να υποστηρίξουμε τις ε, ε, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, των Ρώμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω να ακούσω για να καταλάβω καλύτερα πώς έχει η κατάσταση. Ξεκινάμε το πρώτο πάνελ. Διδάγματα της πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού πλαισίου για, την, για τις, ε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών ένταξης στον Ρωμά. Πρώτοι ορογορητές και όποιοι θέλουν να θέσουν ερωτήσεις μπορούν να το κάνουν μετά. Καλωσορίζουμε τον κύριο Μάρτον Ρόβιντ, υπεύθυνο έρευνα και πολιτική στη στην, ε, στο ίδρυμα, στην γραμματεία του ιδρύματο για την δεκαετία της ένταξη των Ρωμά. Ένα ίδρυμα των ζητημάτων των μειονοτήτων στην, Διεθνή Ακαδημία, στην Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών. Έχετε το λόγο κύριε Ρόβιντ. Και ευχαριστώ και εγώ και για την πρόσκληση και την οργάνωση αυτού του σημαντικού πάνελ. Θα σας συνοψίσω τα ευρήματα της έκθεσης που ανέφερε η κυρία Γκάντσα. Έχω και εγώ και μια παρουσίαση PowerPoint, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Με δύο λόγια θα σας πω πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη συμμόρφωση με το πλαίσιο και τα αποτελέσματα κατόπιν της παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών. Θα σας πω δύο λόγια για το μέλλον του πλαισίου της Ένωσης και το πιθανό ρόλο του Κοινοβουλίου. Επόμενη διαφάνεια. Η εικόνα είναι πολύ σύνθετη. Να σας πω εντάχει ότι για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την διεθνή συμμόρφωση, την αξιολόγηση των πληροφοριών και την, ε, την ε, συλλογή πληροφοριών και την αξιολόγηση, πρέπει να έχουμε μια σειρά πράξεων που σχηματικά περιγράφονται εδώ. Βλέπουμε ότι το σύνθετο, τα σύνθετα αυτά συστήματα υπάρχουν στη Σύμβαση για την Εξάλληψη κάθε μορφή διακρίσεων κατά των γυναικών τον ΙΠΑ, στο, στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Στην περίπτωση των Ρωμά έχουμε δύο ατελή συστήματα. Είναι η δεκαετία της ένταξης των Ρωμά και το πλαίσιο της Ένωσης που συζητούμε τώρα. Στην δεύτερη περίπτωση αυτό που λείπει είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, ε, υποχρεωτικές έκθεσεις πρόοδου ανακράτως, ε, αναθεώρηση των σκιωδών εκθέσεων και ειδικέ συστάσεις αναχώρα. <coughs> Επόμενη διαφάνεια. Αυτό που κάναμε στο πιλωτικό έτος ε, σκιώδους εκθέσεως που έγινε από τις πρωτοβουλίες Ρωμά και από την εκμετάλλευση των πόρων της Ένωσης για τα προγράμματα Ρωμά είναι ότι μετά από ανοιχτή πρόσκληση κάνουμε επιλογή συμμαχίες κοινωνίας των πολιτών από 8 χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Μακεδονία, Ρωμανία, Σλοβακία και Ισπανία. Δώσαμε ένα πλαίσιο, template ε, με, αυστήρα, με αυστηρή επαγγελματική εξέταση και αυτές οι ευρείες συμμαχίες παρακολούθησαν τις επιπτώσεις επιτόπου των μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσει το 12 και ειδικά για του Ρωμά και γενικά διοικητικά μέτρα. Στην είσοδο βρήκατε και μία συνοπτική έκθεση, υπάρχουν και online. Στην άλλη διαφάνεια μπορεί να δείτε πώς μοιάζουν. Μπορεί να κα, κατεβάσετε την έκθεση αυτή άμα θέλετε και από το ίντερνετ. Αποτελέσματα. Βρήκαμε η κοινωνία των πολιτών δηλαδή βρήκε θετικά μέτρα από τις στρατηγικές και γενικά θετικά μέτρα ευρεία πολιτική που ήταν θετικά για του πληθυσμού των Ρωμά. Τα καλύτερα ευρήματα είναι ότι υπάρχουν πολλά θετικά μέτρα αλλά που δεν έχουν σχεδιαστεί επαρκώ ή δεν έχουν υλοποιηθεί επαρκώ και εδώ ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών είναι κρίσιμο. Να δείχνει τα κενά. Επίση υπάρχουν αρνητικά μέτρα των στρατηγικών και των βασικών μέτρων πολιτικής. Επόμενη διαφάνεια. Δεν θα σας πω τα στοιχεία αυτά, διότι έχω περιορισμένο χρόνο. Δύο-τρία μόνο για τις χώρες που, διάφορες χώρες για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Μία, ένα επιτυχές μέτρο στην Τσεχία είναι τα προγράμματα παιδαγωγικής βοήθειας στο Ρωμά. Στη Ουγγαρία υπάρχουν, στη Ρουμανία υπάρχει μια πολύ καλή θετική δράση για γυμνάσια και πανεπιστήμια. Στην επόμενη διαβάνεια βλέπετε γενικά μέτρα που, που ωφέλησαν τους Ρωμά στην Ισπανία. Το δίκτυο κατά των διακρίσεων αντένα. Τώρα να δούμε τα μέτρα που θα μπορούσαν να είναι καλά, αλλά που το 12 δεν εφαρμόστηκαν σωστά. Στην Ουγγαρία. Η κοινωνία, τα προγράμματα κοινωνικών λειτουργών βοήθεια των γυναικών Ρωμά. Πρέπει να βελτιωθούν η επιλογή και η κατάρτιση. Στη Ρουμανία υπάρχουν προγράμματα βοήθεια στην ανασύντηση εργασία που μπορούν να αυξηθούν και να βελτιωθούν. Επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε ότι δυστυχώ κάποια από, τα, από τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν το 2012 στις στρατηγικές δεν ήταν θετικές για την κοινότητα Ρωμά. Στην Ουγγαρία το δημόσιο πρόγραμμα απασχόλησης δεν είναι καλό γιατί δεν παρέχει πρόσβαση στην πρωτογενή αγορά εργασία, όχι μόνο στη Μακεδονία αλλά και αλλού. Η, υποδομ... ανάπτυξη των υποδομών δεν αντιμετωπίζουν την... Ε, το διαχωρισμό κατοικιών. Ενώ στην ε, Σλοβακία δεν υπάρχει καμία προπαρασκευαστική τάξη για του Ρωμά. Επόμενη διαφάνεια. Γενικά μέτρα που ήταν αρνητικά για του Ρωμά. Στην Τσεχία έγινε μια μεταρρύθμιση της, ε, του, της κοινωνικής, ε, του κοινωνικού συστήματος που, που μείωσε την, ε, τα επιδόματα των Ρωμά. Στην Ισπανία υπήρξε μείωση των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων για κοινωνικά μειονεκτικούς μαθητές που, ήταν κυρίως, που έπληξε κυρίως του, τους Ρωμά. Συνολικά, Θέλω να το τέσσερα διδάγματα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο βάσει των αποτελέσματων. Ένα σημαντικό, το τονίσαμε, χρειαζόμαστε πιο ουσιαστική συμμετοχή των Ρωμά. Πρέπει να σκεφτούν τι βλέπουν επί τόπου και ε, αυτά πρέπει να τα σκεφτούν οι εθνικοί και οι διεθνείς διαμορφωτές πολιτικής. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε. Οι βασικές γενικές πολιτικές δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις στοχοθετημένες, στα στοχοθετημένα μέτρα. Επίσης, είναι σημαντικό να χτυπήσουμε την προκατάληψη κατά τον Ρωμά στην εκπαίδευση, στα μέσα, στο ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Δηλαδή οι στρατηγικές δεν δουλεύουν αν δεν υποστηριχθούν από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Τέλος, βρήκαμε ότι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην ένταξη των Ρωμά δεν είναι επαρκής οι επιχειρήσει και οι εταιρείε μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα στον τομέα αυτό. Επόμενη διαφάνεια. Πώς θα αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο μετά τα ευρήματά μα. Υπογραμμίζω τέσσερα πράγματα εκ νέου. Πρώτον, ένα τεχνικό θέμα. Είναι σημαντικό να απλοποιηθεί η παρακολούθηση και, και ο απολογισμός του πλαισίου. Αυτό νομίζω ότι γίνεται και θα εξελιχθεί. Επίσης, προτείνουμε να δημιουργηθούν ομάδες ε, εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της Task Force των ΕΟΜΑ και τα εθνικά σημεία επαφής. Δεν είναι επαρκώς ισχυρά. Ε, ε, επίσης προτείνουμε να υπάρξει εξωτερική εξέταση της χρήσης των ευρωπαϊκών πόλων και το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα κερδίσει από μια παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του hate speech. Τελευταία διαφάνεια, να τονίσω κάποια σημεία για τον πιθανό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει έκθεση προόδου από την Επιτροπή με πολύ πιο λεπτομεριακές συστάσεις και αξιολογήσεις αναχώρα. Επίσης, το Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει την υποστήριξη της παρακολούθησης από την κοινωνία πολιτών της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών ένταξη των Ρωμά. Τρίτον, συστήνουμε στο Κοινοβούλιο να πάρει ηγετικό ρόλο υιοθετώντα ένα ψηφίσμα που καταδικάζει κάθε, κάθε έκφραση, εκδήλωση ρατσισμού κατά τον Ρωμά στα κράτη-μέλη και να αναγνωρίσει τον αντιτσιγκανισμό ισότιμα ως μια καταγγελία ισότιμη με τον αντισημιτισμό. Και τέλος να υποστηρίξει την πρόταση σύστασης ε, του Συμβουλίου από την Επιτροπή για την ένταξη του ΕΡΜΑ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και όλας ε, που μιλήσατε εντός του χρόνου σας για να έχουμε ε, χρόνο και για την περαιτέρω συζήτηση. Θα πρέπει στο μεταξύ να ακούσουμε τις παρουσιάσεις δύο άλλων προσκεκλημένων. Πρώτα του κυρίου Γιούλιους Ρόστας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 αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή μου να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ σήμερα για ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο είναι η πολιτική των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω και να θέσω μια ερώτηση. Καταρχήν θα αναφερθώ στη συμμετοχή των Ρώμα. Θα αναφερθώ στο θέμα τη καταπολέμηση ε, των διακρίσεων ε, θα αναφερθώ ε, στην εκπαίδευση και φυσικά το καυτό ερώτημα τι πρέπει να γίνει. Όσον αφορά τη συμμετοχή των Ρωμά, πιστεύουμε ότι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν υπάρχει κάποιος επίσημος μηχανισμός που να διασφαλίζει τη συμμετοχή των Ρωμά σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει κυρίως μέσω μηχανισμούς εκπροσώπησης εθνικών μειονοτήτων. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρώμα ξεπερνούν ε, τα ε, θέματα των εθνικών μειονοτήτων. Για παράδειγμα, ε, ανακούφιση από τη φτώχεια και άλλα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με τέτοιους μηχανισμούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την πλατφόρμα για τους Ρωμά που δεν ε, ξεκινάει διάλογο με τους Ρωμά συνήθως. Στις συναντήσεις δεν συμμετέχουν ε, Ρωμά ακτιβιστές. Πώς λοιπόν ε, να συμμετέχουν, πώς να συμμετέχουν οι Ρωμά σε μια τέτοια πλατφόρμα. Έχοντας λοιπόν κατά νου αυτή την εικόνα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, έχουμε μάθει τίποτα από το παρελθόν από εθνικές στρατηγικές προενταξιακές, για παράδειγμα. Ένα σύνθημα της δεκαετίας ε, της ένταξης των Ρωμά έλεγε ότι η συμμετοχή των Ρώμα ε, θα είναι αποφασιστικής ε, σημασίας. Πρέπει όμως να ξεφύγουμε από τα συνθήματα και να διασφαλίσουμε έναν πραγματικό διάλογο με τους Ρωμά. Εμένα μου φαίνεται ότι ήδη από τα πρώτα βήματα στη διαδικασία αυτή από την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την υποβολή των εθνικών στρατηγικών από τα κράτη-μέλη και κατά την εφαρμογή δεν έχει ληφθεί υπόψη επαρκώς η συμμετοχή των Ρωμά ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από τα κράτη-μέλη. Και έχουμε το όλο θέμα των διακρίσεων. Πριν λίγες μέρες ε, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέφερε ότι κοινωνική ένταξη των Ρωμά δεν θα μπορέσει να γίνει στην πραγματικότητα εάν δεν ε, καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις εις βάρος τους και την νοοτροπία κατά των Ρωμά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνουν όλα αυτά πέρα από την νομοθεσία ε, κατά των διακρίσεων. Συνήθως ο νόμος κατά των διακρίσεων ε, λειτουργεί αρνητικά σε περίπτωση παραβίασης δηλαδή ενώ πρέπει με θετικό τρόπο να προωθήσουμε την ποιότητα στους χώρους αυτούς και θα πρέπει να προωθήσουμε την ισότητα και να αποτρέψουμε τις της διακρίσεις και υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού πλαισίου ε, και για τα ε, και των εθνικών στρατηγικών ε, και είναι η απομόνωση των Ρώμα. Όσους πόρους και αν επενδύσουμε, εάν δεν εξαλείψουμε αυτά τα σημαντικά εμπόδια δεν θα πετύχουμε αποτελέσματα και τελικά θα κατηγορούμε τους Ρώμα για την, για την ε, αποτυχία των πολιτικών. Επίσης θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση ε, σχετικά με την ε, οδηγία κατά των εθνοτικών, για την ισότητα των για την ισότητα. δεν να αναφέρεται εκεί πουθενά το θέμα του απομονωτισμού. Ε, δεν απαγορεύεται ο φυλετικός διαχωρισμός ε, και γι' αυτό ε, δεν μας κάνει εντύπωση που πολλοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις για να γίνει διαχωρισμός των παιδιών Ρωμά στην εκπαίδευση. Και γιατί συμβάνει κάτι τέτοιο. Ο μηχανισμός λειτουργεί αρκετά εύκολα διότι όταν θέλουμε να εξισορροπήσουμε την αποτελεσματικότητα και τον αριθμό των ε, ε, εποφελουμένων σε μια σειρά προγραμμάτων, ε, ξεχνάμε συνήθως τα δικαιώματα των παιδιών. Υπάρχουν διάφορες εκθέσεις πάνω στο θέμα αυτό που μπορείτε να διαβάσετε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε την αποφυγή των διακρίσεων σπονδυλική στήλη των εθνικών στρατηγικών θα πρέπει να στείλετε ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το θέμα αυτό και συνδέεται με τα δύο πρώτα θέματα και ε, η δημιουργία ε, γνώσης για τους Ρωμά. Πού, ε, πού ακριβώς βασίζουμε τις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Μιλώ για γνώση πέρα από τις στατιστικές. Οι στατιστικές είναι σημαντικές, αλλά δεν μας λένε πώς συμβαίνουν τα πράγματα ή γιατί. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε περιορισμένες ε, γνώσεις για τους Ρωμά, κάτι που οδηγεί σε ε, μη επιτυχείς πολιτικές. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Ρωμανικών Σπουδών και ένας τέτοιος φορέας δεν έχει στην ηγεσία του ούτε έναν Ρωμά βρίσκω ότι αυτό είναι τρομερό. Πώς μπορούμε να μιλάμε για συμμετοχή των Ρωμά, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή τους πέρα από τα συνθήματα και να οδηγηθούμε σε πραγματική δημιουργία γνώσης. Ε, πρέπει να μας πούνε τι θέλουν και πώς το θέλουν. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει τώρα. Για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, συμμετοχής των Ρωμά θα πρέπει να υιοθετήσουμε τεχνικές ε, σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ε, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να αναθεωρηθεί ο τρόπος λειτουργίας της ε, πλατφόρμας των Ρωμά, ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν πραγματικό, ένα χρήσιμο διάλογο με τους Ρωμά. Δεν έχει σημασία το ότι οι Ρωμά επικρίνουν τις δουλειές που γίνονται. Θα πρέπει να υπάρχει διάλογος, αλλιώς δεν θα σημειωθεί ποτέ και θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ε, στις ε, κυβερνήσεις ε, ότι η πολιτική μη, μη διάκρισης θα πρέπει να αποτελεί τη, τη βάση της συνεννόησης με τους Ρωμά. Και όσον αφορά τον φιλετικό διαχωρισμό, αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου κατά των διακρίσεων. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για διαχωρισμό των Ρωμά, θα πρέπει να ε, χρηματοδοτούνται σωστά οι πολιτικές και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προς το Εθνικό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στα θέματα αυτά. Η συμμετοχή των Ρωμά θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για έγκριση οποιασδήποτε πρωτοβουλίας χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η συμμετοχική δράση θα πρέπει να βελτιώσουμε τις γνώσεις για τους Ρωμά ως προϋπόθεση για ε, την ύπαρξη αποτελεσματικών πολιτικών για τους Ρωμά. Και ε, όσον αφορά τις πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία γνώσης, αναφέρθηκα στο σχετικό ευρωπαϊκό δίκτυο. Τι μπορούν να κάνουν οι ευρωβουλευτές. Εάν θα μπορούσα να επιλέξω ένα θέμα, θα ήταν ε, να ε, αναθέσουν τη διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης έκθεσης ε, σχετικά με την συμμετοχή των Ρώμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι υπάρχει εδώ ήδη από την αρχή σύγκρουση συμφερόντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση για να μπορέσει να αναθέσει μια τέτοια ανεξάρτητη μελέτη. Ο τρόπος που ταπανώνται τα χρήματα δεν είναι ε, ευθύνη μόνο των εθνικών κυβερνήσεων, είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρώστας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ επίσης που κρατήσατε και το χρονοδιάγραμμα, διότι έχουμε και μία τρίτη μαρτυρία και μία τρίτη παρουσίαση από τον κυρία Λίνα Παπαμιχαλοπούλου από την Αγαμά ΔΕΛΤΑ Justice συντονίστρια πολιτικών κατά των διακρίσεων και των Ρωμά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι μάρτυρας, είμαι κατηγορούμενη από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Θα περιοριστώ λοιπόν σε κάποια πολύ βασικά θέματα, θέματα αρχής και δεν θα σπαταλήσω χρόνο μπαίνοντας σε λεπτομέρειες και επιμέρους ζητήματα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν δεν ε, θα σας ωρεοποιήσουμε τα πράγματα από ό,τι ακούσαμε από τις ε, μαρτυρίες των συναδέλφων και από τις ε, παρουσιάσεις και από τις εισηγήσεις και επί τη ευκαιρία να σα ευχαριστήσω που με καλέσατε. Βλέπουμε ότι δεν είναι μυστικό, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την ένταξη των Ρωμά. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα. Βρισκόμαστε μόνο δύο χρόνια ε, δύο χρόνια από την έναρξη του πλαισίου που θα τελειώσει το 2020. Ας τα πιάσουμε λοιπόν από εκεί τα πράγματα. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε αυτά τα δύο χρόνια. Θετικά είναι τα εξή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα κράτη-μέλη είτε έχουν μια εθνική στρατηγική είτε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων. Εκτός από τη Μάλτα. Όμως και πάλι να πω προ υπεράσπιση ε, της ε, μάλτα ότι μα έστειλαν μία επιστολή στην οποία συμπεριέλαβαν μία αξιολόγηση των ε, μέτρων σε περίπτωση που έχουν πληθυσμό Ρωμά. Παρότι λοιπόν δεν υπάρχει κάποια έκθεση προόδου, μας έστειλαν αυτήν την στρατηγική. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πολιτικά όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ένταξη των Ρώμων. όχι μόνο πολιτικά, αλλά και η κοινωνία το έχει αναγνωρίσει αυτό. Υπάρχει λοιπόν ευθύνη και αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, ε, κάνουμε εκθέσεις και δίνουμε αναφορές στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μία φορά το χρόνο για την πρόοδο αυτή. Μέχρι τώρα έχουν γίνει δύο τέτοιες εκθέσεις. Η πρώτη από αυτές που εκδόθηκε το 2012 αφορούσε την αξιολόγηση των στρατηγικών, των σχεδίων δράσης, των μέτρων πολιτικής ολοκλήρωσης που μας έχουν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη. Και ούτε εδώ βέβαια δεν θα εκπλαγεί κανείς ότι η εικόνα δεν ήταν ρόδινη. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Ωστόσο, στην έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε επίσης και ένα υπηρεσιακό έγγραφο εργασία όπου εντοπίστηκαν οι αδυναμίε που είχαν όλε αυτέ οι στρατηγικέ. Δημοσιεύτηκε λοιπόν και δημόσια και μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Για κάθε ένα κράτος μέλο έχουν εντοπιστεί αδυναμίε. Και αυτές τι αδυναμίες τι έχουμε καταγράψει. Ταυτόχρονα εντοπίσαμε και αδυναμίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αυτές οι στρατηγικές, αυτές οι στρατηγικές χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα. Η Λίβια, η κυρία Γκόντς και οι συνάδελφοι με εδώ δεν είπαν κάτι το καινούριο και είναι συνάδελφοι και συνεργάτες μου εκείνοι που προανέφερα. Υπάρχει πρόβλημα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε εντοπίσει ο, επίσης ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Λείπει η φωνή των Ρωμά, παρότι όλα αυτά τα μέτρα είναι για εκείνους. Έχουμε επίσης εντοπίσει το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης χαμηλή, διότι υπάρχουν διοικητικά προβλήματα, διότι υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης και έχουν εντοπιστεί λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα και αναφέρονται στην ε, έκθεσή μας. Ωστόσο, να σημειώσω ότι έχουμε και άλλη μία επιτυχία και αυτή είναι το ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, ορίσει εθνικά σημεία επαφής. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα εθνικά σημεία επαφής από ό,τι είδαμε δεν έχουν τη δυνατότητα συντονισμού, δεν έχουν πόρους, δεν έχουν προσωπικό, όμως ασκούμε πίεση. Και εδώ μπαίνουμε και εμείς. Εμείς έχουμε δημιουργήσει αυτά τα εθνικά σημεία επαφής, ήμασταν εκεί, τους ασκήσαμε όση πίεση μπορούσαμε, φυσικά εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων μας. Υπάρχει όμως κοινή ευθύνη Κοινή ευθύνη για την Κομισιόν, για το Συμβούλιο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο ένα θεσμικό όργανο. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία και με την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε λάβει σκιώδει εκθέσεις από όσου, όλους όσους επιθυμούσαν να μα τις στείλουν και δεν περιοριζόμαστε ε, στο, στο ποιος θα μας στέλνει Είμαστε πάντα ανοιχτοί για συνεργασίε. και μάλιστα να σας πω και ότι ένας ε, Ούγγρος γιατρός μας έστειλε εκείνο μία έκθεση. Ένας Ούγγρος γιατρός ο οποίος ε, ασχολείται με ένα πρόγραμμα εμβολιασμού. Δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε ότι θέλουμε βοήθεια. Φυσικά θέλουμε βοήθεια. Επίσης, φέτος, πέραν όλων αυτών, έχουμε προτείνει μία πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου. Διότι έχουμε εντοπίσει όλα αυτά τα προβλήματα και μια ήπια νομοθεσία έχει καλές ευκαιρίες να περάσει. Μια που μιλάμε και όλες για ομοφωνία διότι σύμφωνα με το άρθρο 19,1 παράγραφος 1 της συνθήκης χρειάζεται ομοφωνία. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική πίεση και η μόνη πολιτική πίεση που είχε ασκηθεί ποτέ στα κράτη-μέλη ήταν από, τις, ε, από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Οτιδήποτε άλλο. Στρατηγικές συστάσεις επιτροπής, αποφάσεις επιτροπής δεν έχουν καμία άμεση ε, πολιτική πίεση στις, ε, στα κράτη-μέλη. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου όμως έχουν. Η καταπολέμηση των διακρίσεων, η αποτελεσματική καταπολέμησή τους είναι επίσης σε μία από τις κύριες συστάσεις μας στην πρώτη έκθεση και προϋπόθεση για οποιαδήποτε επιτυχημένη στρατηγική. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα με όλα όσα υπόθηκαν να ξεκαθαρίσω όμως ότι δεν είναι μόνο θέμα της Επιτροπής ή το τι θα μπορούσε ή δεν μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Ξέρουμε ήδη. Έχουμε δημοσιεύσει εκθέσεις. Συνεργαζόμαστε με την Γραμματεία για την επόμενη έκθεση. Διότι η, η επόμενη έκθεση το 2014 θα αφορά και τους τέσσερις πυλώνες και την, την πρόοδο γενικότερα. Θα γίνει εξελόγηση των στρατηγικών και θα εντοπιστούν και οι, διαρθρωτικές, οι ελλείψεις στις διαρθρωτικές προϋποθέσεις. Το 2014 λοιπόν αυτή η έκθεση θα καλύψει αυτούς τους τομείς και αυτή τη χρονική περίοδο. Αυτό κάνουμε λοιπόν, έχουμε κάνει ορισμένε συστάσεις για την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και πιέζουμε πάλι για συγκριτική αξιολόγηση των κονδυλίων αυτών. Εντάξει, δεν θα τα σχολιάσω αυτά διότι δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα, όμως ελπίζουμε να γίνει αυτό. Και αυτά είχα να πω. Είμαι ανοιχτή σε κάθε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους σας. Τώρα, όσοι θέλουν να μιλήσουν μπορούν να ζητήσουν το λόγο. Δύο-τρία λεπτά το πολύ, όχι παραπάνω, για να έχουμε λίγο χρόνο και για απαντήσεις πριν ξεκινήσουμε το δεύτερο πάνελ. Ο κύριος Κλέης ζήτησε το λόγο. Θα είμαι σύντομο, πρόεδρε. Κάθε φορά που ασχολούμαστε με τα θέματα των Ρωμά στο Κοινοβούλιο, διαπιστώνω ότι υπάρχει κάτι που δεν θίγεται της προσωπικής ευθύνης του καθενός. της βοήθειας που οι κοινότητες πρέπει να προσπαθήσουν να συμβάλλουν. Δεν πρέπει αποκριστικά να μιλάμε για Ρωμά ως θύματα. Και δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι έτσι. Θα έπρεπε να τολμήσουμε να μιλούμε για προβλήματα που δεν έχουμε θίξει ακόμα όταν συζητούμε τα ζητήματα Ρωμά. Φερρυπίν. Ξέρουμε ότι στις κοινότητες Ρωμά πολλά παιδιά δεν πάνε σχολείο. Επίσης, μεταξύ των Ρωμά υπάρχει υψηλή εγκληματικότητα. Ο καθηγητής Ντίνα Ζίγκλ από το Βίλεμ Πομπ Ινστιτούτο της ε, Ουτρίχτης που κάνει έρευνα για θέματα εγκληματικότητας και κάνει μία μελέτη πέρυσι για την εγκληματικότητα που λέει ότι όταν αναγγείλαμε ότι θέλουμε να κάνουμε μία μελέτη για το ζήτημα αυτό, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά εμπόδια που είχαν θέσει οι ΜΚΟ όπου εκπροσωπούσαν Ρωμά, θεωρώντας ότι πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. υπάρχει στην κοινότητα των Ρωμά μια ομάδα ε, κλεφτών σπιτιών Ρωμά, δεν είναι όλοι Ρωμά αλλά είναι κυρίως Ρωμά, που ε, λιμένονται την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά κράτη-μέλη. Αυτά... Σε ευχαριστώ κύριος Μπρόνς. Um, if there's anything worse than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 μία ηθελημένη κατηγορία ενάντια ενός ε, λαού ε, ε, διαφέρει από μία μη Ε, Για ποια μιλώ, για ποια κατηγορία μιλώ. Είναι όχι απλά φρικτή, αλλά είναι και πολύ λεπτή. Οι Ρώμα θεωρούνται άνθρωποι θύματα που δεν έχουν κάνει τίποτα όμως για να βοηθήσουν σε αυτούς τους θεωρούνται άνθρωποι που δεν, ε, μπορούν, που δεν έχουν ευθύνη για ε, τα προβλήματά τους ε, αλλά και άνθρωποι που δεν που δεν, έχουν, δεν θεωρούνται ούτε υπεύθυνοι για τις επιτυχίες τους. δηλαδή είναι άλλοι υπεύθυνοι για τη μοίρα τους. δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο ταπεινωτικό για κάποιον. καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να κάνουμε γενικεύσεις, ιδιαίτερα για λαούς, αλλά αλλά μάλλον στους εαυτούς μας ε, θα πρέπει να επιβάλλουμε να μην ε, ε, χρησιμοποιούμε γενικεύσεις για άτομα. Τι γενικεύσεις μπορούμε να κάνουμε και τι ήδη έχουν γίνει σήμερα το απόγευμα σχετικά με την πολύ κακή οικονομική κατάστασή τους και τις κακές κοινωνικές τους συνθήκες. Μπορούν να αλλάξουν από άλλους για τους ανθρώπους αυτούς. Πιθανότατα ναι, αλλά όχι χωρίς την ε, συγκατάθεσή τους και μια απόλυτη αλλαγή του τρόπου ζωής, δηλαδή μια προσπάθεια να επιβληθεί άλλος τρόπος ζωής σε έναν λαό, ε, δεν ε, ενδείκνυται. Θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες, ιδιαίτερα για τα παιδιά τους, αλλά βέβαια η συνεργασία εξορισμού απαιτεί συγκατάθεση και είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί μια τέτοια πολιτική στους ανθρώπους αυτούς. Όσον αφορά λοιπόν αυτές τις γενικεύσεις, μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις ε, για τη συμπεριφορά και τις εμπειρίες. Δεν θα αναφερθώ στο ένα χωρίς να αναφερθώ στο άλλο. Ε, μία ακρόαση στη Λίμπε, νομίζω πριν δύο χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, ε, πραγματοποιήθηκε για την εμπορία ανθρώπων και ε, μίλησε και ο αρχηγός της Europol και πολύ προσεκτικά ρώτησα εάν υπάρχει κάποια ομάδα πληθυσμιακή η οποία να εκπροσωπείται δυσανάλογα είτε μεταξύ των ε, εμπόρων ανθρώπων ή μεταξύ των θυμάτων. Και μου απάντησε ότι ε, ε, η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι η Ρωμά. Αντιπροσωπεύονται δυσανάλογα και μεταξύ των εγκληματιών και των θυμάτων. Το να προσποιούμαστε ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα δεν θα επιτρέψει τη λύση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, κάποια ε, οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Ε, σας παρακαλώ, ε, παρακαλώ πείτε μας το όνομά σας και αν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, όσο πιο γρήγορα μας το υποδείξει, τόσο καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι από την Ένωση Ρωμά και Σύντη στις κάτω χώρες. Έχουμε αντιπροσωπεία τεσσάρων ανθρώπων εδώ σήμερα το απόγευμα θα σας παρακαλούσα να ε, εξετάσουμε την ε, διάκριση εις βάρος των ε, Ρωμά στις κάτω χώρες. υπάρχει μια πολιτική για παράδειγμα, εδώ και ε, αρκετά χρόνια ε, δεν μπορεί κανείς να νοικιάσει χώρο να ε, παρκάρει το το τροχόσπιτο και είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε σε σπίτια χωρίζουν οικογένειες, δεν μας δίνουν χρήματα, κρατικές ενισχύσεις. Εξαρτιόμαστε από από το δικό μας εισόδημα ε, και θέλουν να μας εξαφανίσουν. Και η αστυνομία μας παρενοχλεί. Και με ένα σπίτι μου έρχονται να δούνε μήπως ε, πραγματοποιούνται εκεί εγκληματικές δραστηριότητες. Ε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έπρεπε εγώ μόνη μου να πληρώσω για την αλλαγή της κλειδαριάς μου που παραβιάστηκε και είχαμε πολύ κακές εμπειρίες ε, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, ε, έχουμε συλλέξει άρθρα από τον τύπο σχετικά με την Ένωσή μας. Μπορείτε εδώ να τα διαβάσετε. Και ο δήμαρχος ε, της ε, περιοχής μου ε, λέει ότι θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι θέσεις τροχόσπιτων και είναι πρόεδρος της Ένωσης Δήμων των Κάτω Χωρών οπότε ζητάει από όλους τους δημάρχους να ασκήσουν την ίδια πολιτική. Και όσον αφορά τους Ρώμα που έρχονται ε, στις κάτω χώρες ε, χωρίς διαβατήριο και αυτοί αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Ε, πολύ ευχαρίστω να σας ενημερώσω περαιτέρω. Έχουμε άρθρα για ανθρώπους τους οποίους απομάκρυναν από τον τόπο διαβίωσης τους. Θέλουμε λοιπόν να ε, ε, ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο απέναντι στο πρόβλημα και των δυτικών, δυτικοευρωπαίων Ρωμά, όχι μόνο των ανατολικοευρωπαίων. Ε, δεν υπάρχουν όμως αρκετά χρήματα για να λυθούν τα προβλήματά μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως γενικά είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια Έχουμε δει πάρα πολλά περιοριστικά μέτρα στο θέμα της ε, μετανάστευσης εδώ στα κράτη-μέλη. Και πραγματικά αυτό είναι λυπηρό. Και είναι λυπηρό ότι αυτή ακριβώς η ομάδα των Ρωμά ανήκει είναι η ομάδα αυτή που εδώ και πάρα πολλά χρόνια υφίσταται διακρίσεις και έχει να αντιμετωπίσει όλα και ε, αυξανόμενα προβλήματα. Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα, επίσης, ε, λυπάμαι κάθε φορά που ακούω ιστορίες και μαρτυρίες όπως αυτές που ακούσαμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι φυσικά έχουν ε, ε, ευθύνη για τη ζωή τους. Όμως δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε αυτό για τους Ρωμά. Ωραίο είναι να λέμε ότι όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν, στο σχολείο. Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχουν λεωφορεία για να τους πάνε να πάνε αυτά τα παιδιά στα σχολεία που να πηγαίνουν στις περιοχές που ζουν Ρώμα. Τι γίνεται με τις υποδομές που δεν τους επιτρέπουν να ενταχθούν. Και πολλές φορές έχω, ε, άκουσα τώρα στην ε, έκθεση αυτά τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί όσον αφορά την εφαρμογή των ε, μέτρων. Και ανεξάρτητα από αυτά που έχω ακούσει από ορισμένου, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχω ακούσει από ορισμένου από εσά ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι πρέπει να ασχοληθούμε με λύση προβλημάτων, ότι αναφέρθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα σε συγκεκριμένες χώρες και αυτό που πρέπει είναι να πιέσουμε τους αρμόδιους φορείς στις δικές μας χώρες, τουλάχιστον προσπαθώ εγώ να το κάνω αυτό στη δική μου χώρα, να ασχοληθούν επιτέλους με αυτές τις ε, ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Ήδη σε προηγούμενη συζήτηση για την στρατηγική των Ρωμά έχω ξαναπεί ότι έχουμε πάρα πολλές, ε, υπάρχουν πάρα πολλές μειονότητες και υπάρχουν πάρα πολλά ε, πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Και αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι Ρωμά, τότε θα έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόοδο και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλους συναδέλφους να θέλουν το λόγο. Ας κάνουμε... Ας έρθουμε τώρα λοιπόν ε, στην ώρα των απαντήσεων και όσο συντομότερο τόσο το καλύτερο, διότι μας περιμένει και το δεύτερο πάνελ στις 5 παρά τέταρτο. Κύριε Ρόβιντ, έχετε το λόγο. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στις δύο πρώτες παρεμβάσεις. Ε, αυτό που στηρίζω είναι να προχωρήσουμε πέρα από την, ε, από την θεωρήση των Ρωμά ως θύματα και να προχωρήσουμε στην κοινωνική τους ένταξη, να τους θεωρήσουμε πολίτες που έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους. Να... Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτόν τον ε, έτσι, ε, όρο της μόδας, τη χειραφέτηση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όλες οι στρατηγικές πρέπει να έχουν αυτό έντονο αυτό το στοιχείο της χειραφέτησης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρώστας, ευχαριστώ πολύ. Ε... Ως ε, ειδικό για τους Ρωμά, διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο μαθήματα για πολιτικές Ρωμά. Θέλω να σας πω το εξής. Όταν εννοούσα γνώση πέραν των στατιστικών, αυτό εννοούσα. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να νηθούμε πως υπάρχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα μεταξύ των Ρωμά. Αφετέρου, δεν θα σύγκρινα λέγοντας ότι η εγκληματικότητα μεταξύ των Ρωμά είναι υψηλότερη και ποσοτικοποιημένη. Δεν μπορείς να ταυτίσεις δέκα μικροκλοπές με μια μεγάλη υπεξαίρεση στον τραπεζικό τομέα. Τι είναι πιο σημαντικό, δέκα ή μία πράξεις. Αυτό είναι δύσκολο να το συγκρίνεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η εγκληματικότητα δεν είναι θέμα. Αφετέρου. Και ως Ρωμά και ως μελετητής των Ρωμά έρχομαι να σας πω γιατί δεν εφαρμόζεται σωστά ο νόμος από την κυβέρνηση και τις διοκτικές αρχές. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο όταν είναι για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά και όταν οι γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Και εκεί πρέπει να επιβληθεί ο νόμος, γιατί υπάρχει το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση. Δεν είναι απόφαση του, παιδιού, του μπαμπά, του πατέρα να αρνηθεί αυτό το δικαίωμα στο παιδί. Όταν μιλούμε για εφαρμογή του νόμου πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το θέμα αυτό. Και μερικές φορές οι υπηρεσίες των κυβερνήσεων δεν εφαρμόζουν τον νόμο σε άλλους τομείς. Τώρα, καλή η ανταλλαγή ε, απόψε είναι σημαντική. Για την συνένεση η συνένεση απαιτεί δύο. Όταν λείπει μία πλευρά, τι συνένεση να έχει. Προφανώ η εμπορία ανθρώπων είναι ευαίσθητο θέμα και μπορείς εύκολα να το συνδέσεις με του Ρωμά στα στατιστικά γιατί είναι και δράστες και θύματα. Και επανέρχομαι εκ νέου στο πώς εφαρμόζεται ο νόμος. Πολλές φορές και η αστυνομία και οι ιδιοκτικέ αρχέ αρνιούνται να πάνε στι περιοχέ του Ρωμά για να εφαρμόσουν τον νόμο γιατί τους νοιάζει. Είναι τόσο διαφορετικοί που αδιαφορούν για αυτούς. Νοιάζονται μόνο όταν έχουν ε, να κάνουν με την ε, πλειοψηφούσα κοινωνία. Στη διακίνηση να τιμωρηθούν και οι πελάτες, όχι μόνο τα θύματα. Αυτοί που κάνουν τη διακίνηση, αλλά και ο πελάτης. Και συχνά ο πελάτης δεν είναι Ρωμά. Αυτά οι απαντήσει μου. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου πρόεδρος. Thank you. No problem. It's something very common. well, anyway, I will... Ευχαριστώ πολύ. Να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Ρώστας και θα προχωρήσω και ένα βήμα παραπέρα. Ε, δεν είμαι Ρωμά, θα ήμουν περήφανη όμως αν ήμουν. Δεν πιστεύω στις ε, στατιστικές όταν αυτές περιορίζονται σε νούμερα. Πιστεύω σε στατιστικές όταν εκείνες ε, αναλύονται και εξαρτάται πώς ερμηνεύεις μια στατιστική. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για την έκθεση της Europol για την ε, διακίνηση ανθρώπων. Ξέρω όμως που στόχευαν όταν έκαναν την αναλύσή τους. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει άλλη ατζέντα για διακίνηση ανθρώπων, παράδειγμα, προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω. Θα σχολιάσω όμω αυτό που είπε η κυρία Σίπελ και θα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε τα στερεότυπα. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν ενδιαφέρει του Ρωμά η ένταξη. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουν πάρει αποφάσεις για τη ζωή τους, για τα παιδιά τους και γι' αυτό δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε δεν μπορούμε να λέμε ότι εντάξει έχουν πάρει τις αποφάσεις τους και έχουν αναλάβει τις, ευθύνε τις ευθύνες τους. Αυτό είναι το πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα. Αυτό τους έχει δώσει η κοινωνία. Αυτή είναι η ζωή τους. Ζουν τη ζωή τους όπως μπορούν δεδομένων των συνθήκων. Και κάτι άλλο που αναφέρθηκε, όταν μιλάω για διακρίσεις, εννοώ διακρίσεις. Όταν τα παιδιά στην Ουγγαρία ζητιανεύουν στο δρόμο, αν τα παιδιά αυτά είναι Ρωμά, οι γονείς δεν διώκονται ποινικά. Εάν κάποιο άλλο παιδί δεν πάει στο σχολείο, ο διευθυντής παίρνει τηλέφωνο του γονείς και του ρωτάει γιατί. Και αναφέρομαι σε αυτό επειδή το αναφέρατε κι εσείς. Ε, δεν, ε, δεν είναι απαραίτητο να είναι η Ρουμανία, μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν διακρίσει λοιπόν. Όταν εμεί επικοινωνήσαμε με τα εθνικά σημεία επαφή, πολλέ φορέ συν, συνειδητοποιήσαμε ότι όσον αφορά την εκπαίδευση, στη δική μας πρόταση με το Συμβούλιο αναφερόμαστε στην επίτευξη του υποχρεωτικού ε, της υποχρεωτικής ε, διάρκειας της εκπαίδευσης. Στην σύσταση της Επιτροπής αναφέρεται η ελάχιστη διάρκεια. Όχι, η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται ίσα. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς για τις απαντήσεις και για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους καλεσμένους του πάνελ που κατάφεραν να έρθουν εδώ, διότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που ήρθατε και μας εκθέσατε τις απόψεις σας. Τώρα θα δούμε ένα μικρό βίντεο, περίπου 5 λεπτά θα διαρκέσει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να κρατήσει όντως πέντε λεπτά. Θα δούμε.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 Θα μιλήσω σουηδικά τώρα. Eh, eh, Βρίσκω ότι ήταν μια ταινία που δίνει μια εικόνα της Ευρώπης που δεν πιστεύουμε καν ότι υπάρχει. Είναι χρήσιμο να δει κανείς λοιπόν μια τέτοια ταινία και να δει τι συμβαίνει. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων θα ε, πραγματοποιήσει ε, αποστολή εκεί να δούμε τα πράγματα από κοντά. Τώρα λοιπόν που είδαμε την ταινία περνάμε στο δεύτερο πάνελ και θα ήθελα να καλέσω τους τρεις ομιλητές, ε, Μπλάνκα Κόσμα, Φίνα Ρουμπίνα Σεράνο και τον κύριο Γιωάννη Δημητρακόπουλο. Δημητρακόπουλο, συγγνώμη. Ε, παρακαλώ, καθίστε. Okay, thanks. Thanks a lot. Uh, we will now start the second panel. Ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. και θα ακούσουμε πρώτα παρέμβαση της κυρίας Μπλάνκα Κόσμα, εκπρόσωπος ΜΚΟ του Εθνικού Συμβουλίου Υποθέσεων των Ρωμά. Είναι επίσης εμπειρογνώμων ε, ίσων δικαιωμάτων ε, στη Βουταπέστη και πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ρωμά στην ε, δημόσια ζωή. Έχει οργανώσει αρκετά ε, σεμινάρια για την καταπολέμηση της πορνείας ε, και την εμπορία γυναικών Ρωμά. Και έχει δημιουργήσει ε, ένα κέντρο πληροφόρησης για την κοινότητα των Ρωμά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιαρούκο, ε, αξιότιμοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να σας ε, παρουσιάσω την κατάσταση των Ρωμά στην Ουγγαρία. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε και άλλες γυναίκες που έχουν εργαστεί σκληρά επί πολύ καιρό για να πετύχουν βελτίωση της κατάστασης για τους Ρώμα με τη δουλειά τους. Όσον αφορά το πλαίσιο στρατηγικών, πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό που έχει δημιουργηθεί. Διότι εφιστά την προσοχή του κόσμου σε όλο τον κόσμο στο θέμα αυτό, ορίζει στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν και επίσης ε, αναφέρονται οι αρμόδιοι οργανισμοί και δημιουργείται και ένα πλαίσιο παρακολούθησης. Ε, αυτά είναι τα πλέον εκτήματα της στρατηγικής αυτής. Είμαστε επίσης ε, πολύ περήφανοι που το πρόγραμμα αναγνωρίζει ε, την μειονεκτική θέση των γυναικών Ρωμά στην κοινωνία και που αναφέρει δράσεις για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Επίσης αναγνωρίζει τους, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και είναι πρώτη φορά που μια τέτοια στρατηγική καθορίζει τον ρόλο των ε, Μίκιο σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Και ε, ε, αναγνωρίζεται έτσι ο, ρόλος των ΜΚΟ όσον αφορά τους στόχους. 2.000 γυναίκες θα πρέπει να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν στον δημόσιο τομέα. Σήμερα ε, εκπαιδεύονται 500 με 800 γυναίκες ε, και θα είναι πολύ θετικό αν καταφέρουν να προσληφθούν στο δημόσιο τομέα. Εάν αυτό γίνει με επιτυχία και μπορέσουμε να προσλάβουμε 1.000 ή 2.000 ε, γυναίκες Ρωμά στο δημόσιο τομέα, τότε ουσιαστικά θα γράφουμε ιστορία. Υπάρχουν ε, φυσικά και προσδοκίες όσον αφορά το πλαίσιο στρατηγικής και πιστεύω ότι μία στρατηγική είναι ένα μεγάλο ε, έργο ε, το οποίο όμως είναι και κομμένο κεραμένο στα μέτρα των εθνικών κυβερνήσεων. Και για να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση για τις ε, γυναίκες και τα παιδιά των Ρωμά, δεν θα πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο έργο μόνο, ένα μεγάλο πρόγραμμα που να το επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στην εκπαιδευτική πολιτική, τα σχολεία, την πολιτική απασχόληση. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις κύριες εθνικές πολιτικές. Και θα θέλαμε να δούμε και μια στρατηγική που να στοχεύει σε ριζική βελτίωση της εκπαίδευσης για να αντιμετωπίσουμε τα μειονεκτήματα των ανθρώπων αυτών ε, στην εκπαίδευση. Κάθε ε, ευρώ που δίνουμε για την εκπαίδευση ε, ουσιαστικά φέρνει αποτελέσματα στην οικογενειακή πολιτική για την ε, εκπαίδευση των παιδιών. Ε, μπορούμε λοιπόν ε, μέσα στα 15-20 χρόνια να καλύψουμε κενά αιώνων. Η επόμενη στρατηγική, λοιπόν, η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να επιδιώξει να μειώσει τις, τη μειονεκτική, να βελτιώσει τη μειονεκτική θέση. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά και τα παιδιά των νόμων. Δεν θα πρέπει να μειώσουμε την ε, ελάχιστη ηλικία κατάληψης του σχολείου από τα 18 στα 16. Το αντίθετο θα πρέπει να συμβεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο. Θα πρέπει να σταματήσουμε να ε, δημιουργούμε νέους ε, που να μην έχουν δεξιότητες και να μην έχουν καμία ελπίδα στην κοινωνία. Θα πρέπει επίσης ε, να ε, εξετάσουμε και, το, και τις υπηρεσίες υποστήριξης των οικογενειών. Ε, να έχουμε επικοινωνία με μη κυβερνητικές οργανώσεις των Ρωμά και θα πρέπει σε κάθε σχολείο να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των διαφόρων φορέων και να παρακολουθείται η πρόοδος των παιδιών. Και η ε, πόροι θα πρέπει να ε, συνδέονται ακριβώς με αυτή τη συμφωνία και ε, οποιοδήποτε πλεόνασμα στις ενισχύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται και μάλλον οποιαδήποτε επιπλέον ενίσχυση θα πρέπει να προποθέτει την καλή πρόοδο του παιδιού. Σήμερα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις των Ρωμά δεν έχουν καμία πρόσβαση στα σχολεία. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο τύπο συνεργασία με τα σχολεία. Δεν ε, βλέπουμε όμως από μέσα τις εγκαταστάσεις των σχολείων. Εμείς και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα σχολεία και να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η πρόοδος των παιδιών ε, εκ των έσω. Έτσι φτάνω σε στο πρόγραμμα του 2009 για τις γυναίκες ε, είχαμε κάποιες ανησυχίες σχετικά με το αν αυτό θα έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ε, για τις θέσεις απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Αν καταφέρουμε όμως να αλλάξουμε την πολιτική ε, της εκπαίδευσης θα υπάρξουν πολλές δουλειές στον δημόσιο τομέα για τις γυναίκες αυτές. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία. Και δεν μιλώ για τα δημοτικά μόνο. Μιλώ και για σχολεία ενηλίκων Θα πρέπει λοιπόν ε, να αλλάξει η διαπίστευση των σχολείων, ε, τα σχολεία να μπορούν ε, να δέχονται και ενήλικες. Και θα πρέπει και σε λύκια να έχουν πρόσβαση τα παιδιά των Ρωμά. σήμερα στα βορειοδυτικά της Ουγγαρίας, όπου γνωρίζω πως έχει η κατάσταση, τα παιδιά δεν βρίσκουν λύκια να εγγραφούν. Τα σχολεία που έχουν καλή φήμη δεν ε, δέχονται Ρωμά. Θα πρέπει τα σχολεία, τα καλά σχολεία να έχουν ε, ε, παρατήματα σε χωριά, σε μικρές πόλεις και αυτό θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Επίσης θα πρέπει να δούμε πού Υπάρχουν και νέες θέσεις απασχόλησης. Ε, πολλές γυναίκε Ρωμά σήμερα εργάζονται στον τομέα τη υγεία. Είναι χαμηλή αμοιβή και παρέχουν πολύ καλή δουλειά. γυναίκε ε, που παρέχουν κατάρτιση ε, για νοσοκόμε κλπ. θα πρέπει να δέχονται περισσότερε γυναίκε Ρωμά. ώστε να μπορούν και αυτές να αποκτούν επαγγελματικές δεξιώσεις, δεξιότητες. Αλλιώς ε, οι νέοι των Ρωμά δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά και θα έχουμε μακροπρόθεσμη ανεργία. Αυτή... Αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα της κοινότητας των Ρωμά, διότι όσα και να μάθει κανείς, ακόμα και αν ε, σπουδάζει κανείς ε, σε πανεπιστήμιο ή πηγαίνει στο Λύκειο, ε, συχνά δεν βρίσκει κανείς δουλειά. Πολλοί άνθρωποι στην Ουγγαρία ή και στις δυτικές χώρες ε, δουλεύουν σε χειρονακτικές δουλειές, δουλεύουν ως καθαριστές, διότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά που να αντιστοιχεί στις ε, ειδικότητε τους. Η πολιτική απασχόλησης θα πρέπει να προβλέπει θετικές διακρίσεις ώστε να βρίσκονται θέσεις πρακτικής, απασχόλησης, πρακτικής ε, άσκησης ε, και θέσεις εργασίας ε, για τους Ρώμα. Η μακροπρόθεσμη ανεργία είναι πάρα πολύ δαπανηρή και για τον προϋπολογισμό, αλλά γενικά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σχολιάσω ε, κάτι για εκείνους που δουλεύουν και τα βλέπουν αυτά στην πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να βλέπω καθημερινά ε, Ρωμά και να ακούω εμπειρίες. Τα χειρότε, οι χειρότερες εμπειρίες που έχω δει είναι περιπτώσεις νέων γυναικών Ρωμά που παρόλη την εκπαίδευση, ή την κατάρτισή τους δεν μπορούσαν να βρουν κάποια ε, θέση εργασίας. Πιστεύω πως η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης για τους ε, Ρωμά πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό. Μου μένουν τώρα μερικά λεπτά και θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στην κατάσταση των γυναικών ε, Ρωμά όσον αφορά την απασχόληση. Δυστυχώς, οι εμπειρίες μου είναι πάρα πολύ δυσάρεστες. Οι γυναίκες ε, Ρωμά στην Ουγγαρία απασχολούνται μόνο κατά το 13% σε κατάλληλες θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις νομικές προδιαγραφές και ακόμα και αυτό το 13% που εργάζεται εργάζεται κάτω από άσχημες συνθήκες ε, με το βασικό μισθό, απειλούνται ε, με απόλυση γι' αυτό οι γυναίκες αυτές ε, χρειάζεται πολλές φορές να κάνουν δύο ή τρεις δουλειές ταυτόχρονα έτσι ώστε να καταφέρουν να βγουν από τη φτώχεια και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Έχουν λοιπόν επίσημα μία δουλειά, αλλά πρέπει να κάνουν και άλλες δύο. Οι καθαρίστριες στην Ουγγαρία που δουλεύουν στην, ε, στο Υπουργείο Οικονομικών ε, της ε, Ουγγαρίας μας λένε ότι οι συνθήκες εργασίας τους είναι πάρα πολύ άσχημες, ότι γίνονται κρατήσεις, ότι δεν τους ε, δίνονται οι επιστροφές σε φόρου που δικαιούνται και ότι αυτές ε, πάντα κατακρατούνται από τους εργοδότες παρότι οι γυναίκες αυτές αναγκάζονται να υπογράψουν ε, ότι έλαβαν τα χρήματα αυτά. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι γίνεται με το υπόλοιπο 17% που δουλεύουν στην παραοικονομία. Πόσο ασφαλής είναι η εργασία τους, πόσο εύκολα απολύονται. Αυτές οι γυναίκες είναι εκτιθυμένες σε πολύ αρνητικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια της ε, ζωής τους και έχω πάρα πολλές ε, ιστορίες να σας πω. Για παράδειγμα, μία φορά μια γυναίκα χρειάστηκε να λείψει για να πάει σε μια κηδεία και την επόμενη μέρα χάσε τη δουλειά της. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ε, και γυναικών που δουλεύουν με συμβάσεις έργου και δεν παίρνουν το μισθό που τους ε, αναλογεί σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει. Για να μην μιλήσω και για τους ε, χιλιάδες που απασχολούνται στον κατασκευαστικό τομέα. Στην Ουγγαρία πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να βγάλουν έξτρα κέρδος. Οι, εταιρείες, οι οποίες εταιρείες δεν τους πληρώνουν όσο θα έπρεπε και το δυστυχέ αυτές τις, τις περιπτώσεις είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καν το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης και σε περίπτωση που πεθάνουν, για παράδειγμα, τα μέλη της οικογένειάς τους ή οι κληρονόμοι τους δεν έχουν το δικαίωμα κοινωνικών παροχών και αυτό το φαινόμενο ολοένα και εντείνεται. Η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη. Επίσης, να αναφερθώ και λίγο στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στην ε, υποστήριξη της ε, κοινωνίας των πολιτών αν έχω το χρόνο. Δεν έχω πολύ χρόνο από ό,τι πληροφορούμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε και το ζήτημα της ε, στήριξης από την κοινωνία των πολιτών, γιατί πάρα πολλοί νέοι Ρωμά δεν μπορούν να βρουν δουλειά παρά μόνο μέσα από μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή από διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτές οι οργανώσεις δεν έχουν κονδύλια, δεν έχουν ίδιους πόρους και πολλές φορές οι, οι Ρωμά δεν, μπορούν καν να... δεν είναι καν στη θέση να ζητήσουν τις κοινωνικές αυτές παροχές. και πολλές φορές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια που διατίθενται για τα προγράμματα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που εργάζονται στα προγράμματα αυτά για τους Ρωμά, εργάζονται όμως και δεν συνεργάζονται με τους Ρωμά και αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολη την έβρεση εργασίας και η εμπειρία μας δυστυχώ είναι άσχημη. Πολλές φορές ακόμα και αν ε, βρουν κάποια θέση εργασίας σε ένα έργο, μόλις τελειώσει αυτό το έργο τότε χάνατε και οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί. Δεν μπορούν να βρουν άλλη δουλειά. Και εδώ θα σταματήσω και να σας ευχαριστήσω για το χρόνο. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την εμπειρία σας και την εισήγησή σας. Προχωρούμε. Η κυρία Φίνα Ρούμπιο Σεράνο, εκπρόσωπος ΜΚΟ από την, το Ίδρυμα ΣΟΥΡΤ, της οποίας είναι και πρόεδρος. Είναι μια οργάνωση γυναικών που δημιουργήθηκε το 1993 και βασίζεται στη Βαρκελόνη. Με έχει στόχο την αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ένταξη της έμφυλης διάσταση στο δημόσιο χώρο. Για πάνω από 10 χρόνια η ΦΙΝΑ οργανώνει, συντονίζει προγράμματα για την κοινωνική ένταξη των γυναικών Ρωμά. Έχετε το λόγο. Gracias por la invitación Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μετάσχω στο πάνελ αυτό. Ελπίζουμε ότι η συνεισφορά μας θα είναι χρήσιμη στην ε, συζήτηση και ότι θα μπορέσει να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθήκων ζωής ε, των ε, γυναικών Ρωμά. Το ΣΟΥΤ είναι ένα ίδρυμα που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Έχουμε κάνει μια ευρεία δραστηριοποίηση σε θέματα έρευνας και στην άμεση παρέμβαση στον πληθυσμό των Ρωμά, αλλά και στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Το μεγαλύτερο τμήμα των πληροφοριών που θα σας παρουσιάσω στην εισήγησή μου αποτελεί τμήμα ενός ερευνητικού σχεδίου που έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Daphne Empower, στο οποίο μετέσχουν τέσσερις οργανώσεις από τέσσερις χώρες της Ευρώπης, Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουμανία και Ισπανία. Οι λόγοι που μας οδήγησαν στο ΣΟΥΤ είναι πολλοί. Θα υπογραμμίσω κάποια θέματα που κατά την άποψή μας ε, είναι κεντρική σημασία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βίας των γυναικών κατά των γυναικών εν γέννη και μέσα στις κοινότητες Ρωμά ειδικότερα και που αποτελούν και την αφετηρία του έργου. Ξεκινάμε από μία δήλωση που νομίζω όλοι όσοι είμαστε εδώ παρόντες συμμεριζόμαστε. Η ανδρική βία είναι μια διαδοτική δομική βία που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια και μετά από κοινωνική ανάλυση της βίας κατά των γυναικών είδαμε ότι το φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει κάθε γυναίκα με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από την τάξη, εθνική καταγωγή ή άλλη μορφή ταξινόμησης, κοινωνικής ταξινόμησης. Έτσι, δόθηκε έμφαση στην κοινή εμπειρία όλων των γυναικών απέναντι στην ανδρική βία. Ωστόσο, παρότι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα οριζόντιο φαινόμενο, πιστεύουμε ότι όπως και ο διεθνής φεμινισμός πρέπει να απομακρυνθούμε από μειογενή, από μειογενή λόγο για να καταλάβουμε όχι μόνο τα κοινά χαρακτηριστικά αλλά και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτής της συμπεριφοράς. Οι πατριαρχικές αξίες λοιπόν μπορεί να είναι ίδιες σε όλες τις κοινωνίες, ωστόσο η εκδήλωση, η εκδήλωση τους ποικίλει και προσαρμόζεται στις διαφορετικές ειδικέ κοινοοικονομικές συνθήκες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε τον παραδοσιακό λόγο που ομοιογενοποιεί την πείρα για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να γνωρίσουμε την εμπειρία της εξειδικευμένης βίας κατά των γυναικών. Επόμενη διαφάνεια. Ένα από τα βασικά στοιχεία όταν προσπαθούμε να αναλύσουμε και να καταλάβουμε το φαινόμενο της βίας προέρχεται από τον πολιτισμό, δηλαδή την κουλτούρα. Να καταλάβουμε πώς μια συγκεκριμένη κοινότητα αντιλαμβάνεται, ορίζει, αντιδρά και τοποθετείται εναντί της βίας κατά των γυναικών, πλαισιώνοντας έτσι και το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τη βία, αλλά και τις αξίες, τους κώδικες, τα ορόσημα και τους κανόνες με τους οποίους η κοινωνία συνολικά θέλει να αντιμετωπίσει την βία των γυναικών. Εμείς θεωρούμε σημαντικό να υπογραμμίσουμε τη διαφορά μεταξύ πατριαρχικής, πατριαρχικών, διαφόρων πατριαρχικών κουλτουρών. Αυτές οι κουλτούρες διατρέχουν και τις κοινότητες των Ρωμά παίρνουν ειδικέ μορφές και εκφράζονται με τη δική τους κουλτούρα. Οι εκδηλώσεις αυτές συνιστούν λογικά βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση της αυτότητας των ε, γυναικών Ρωμά και την οργάνωση των κοινοτήτων Ρωμά. Επόμενη διαφάνεια υπογραμμίζουμε μεταξύ των εκδηλώσεων αυτών κάποια από τα βασικά στοιχεία που κατά την άποψή μας επηρεάζουν την ταυτότητα των γυναικών Ρωμά. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία εκφράζεται στο βάρος που έχει κοινωνική συλλογική ταυτότητα η οποία επιβάλλεται με ισχυρό τρόπο στην ατομική ταυτότητα και στις ατομικές ικανότητες, στη συγκεκριμένη περίπτωση των γυναικών Ρωμά έναντι ε, ανδρικής βίας. Άλλο στοιχείο η φυσικοποίηση του σεξουαλικού καταμερισμού της εργασίας που αποτελούν κομμάτι της ε, γυναικείας ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις πατριχικές κοινωνίες, αλλά ιδιαίτερα και στις κοινότητες των Ρωμά που βασίζονται με αυτή την ε, ε, σεξουαλική, το σεξουαλικό καταμερισμό της δουλειά τους. Αποτέλεσμα αυτού, οι, οι γυναίκες Ρωμά είναι οι μόνες υπόφθηνες για την αναπαραγωγή βιολογική, κοινωνική και συναισθηματική της κοινότητας. Αυτή η φυσιοποίηση της ερωτικής, της σεξουαλικής, του σεξουαλικού καταμερισμού της εργασίας θεωρείται ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας των γυναικών Ρωμά. Ως αποτέλεσμα, οι κοινωνικές προσδοκίες για αυτές ορίζονται με βάση την οικιακή ε, δουλειά και αντιστοιχούν σε αυτό το ρόλο με θετικό τρόπο. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η υποταγή στην ανδρική αρχή. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα και από κοινότητα σε κοινότητα ή από γυναίκα σε γυναίκα. Η υποταγή ωστόσο στον άνδρα είναι ένα βασικό στοιχείο στην ε, διαμόρφωση της κοινωνικής οργάνωσης των ε, κοινοτήτων των Ρωμά. Τελευταίο σημείο. Ο σεξουαλικός ρόλος που είναι εξαιρετικά διαδρομένος μέσω των στοιχείων όπως της παρθενίας, βασικό στοιχείο για τις γυναίκες αλλά όχι για τους άνδρες Ρωμά, ο γάμος που θεωρείται ως μία υποχρέωση που αποτελεί στην ουσία συνδυασμό και όχι σύνδεσμο ζωή και η πίστη ένα συστατικό στοιχείο της ε, ύπαρξης του Ρωμά. Αυτά τα στοιχεία είναι κοινά σε όλες τις γυναίκες σχεδόν Ρωμά που ριζώνονται στο πλαίσιο μιας αυστηρής πατριαρχικής ε, ε κουλτούρας που είναι κοινή σε όλους, διασυνδέουν το ρόλο της γυναίκας στην κοινότητα Ρωμά ορίζοντας με απεριοριστικό τρόπο τα μοντέλα άντρα-γυναίκα που αποδέχονται οι κοινότητες αυτές. Επόμενη διαφάνεια. Όταν μιλάμε όμως για την κοινότητα των Ρωμά και τις γυναίκες των Ρωμά θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη διαφορετικότητα. Η ποικιλομορφία αυτή που έχει πολλές αφετηρίες και ξεκινά από διαφορετικές στάσεις που, τρόπου που βιώνει κάποιος την ταυτότητά του ως Ρωμά. Εκπαίδευση, κατάρτιση, αμοιβόμενη εργασία, οικιακή εργασία, κοινωνική συμμετοχή. Πιστεύω ότι κάθε γυναίκα Ρωμά είναι ένας μοναδικός κόσμος. Το είπε και μια γυναίκα που μετήχε σε ένα field work που κάναμε. Σίγουρα η ταυτότητα των ε, γυναικών Ρωμά είναι εξαιρετικά ετερογενής. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία Ρωμά γυναίκα. Υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα και άρα πολύ διαφορετικές εμπειρίε. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτή της ετερογένειας μπορούν να συνεπάρξουν κοινέ διαστάσεις που βιώνουν πάρα πολλέ από αυτές και που σχετίζονται με την ε, λύση συγκεκριμένων ε, παραδοσιακών έμφυλων ρόλων που αποτελούν ε, απαραίτητο τμήμα της ταυτότητας και που ποικίλουν ανάλογα με το διαφορετικό πολιτιστικό, γεωγραφικό και κοινωνικό πλαίσιο κάθε κοινότητας Ρωμά. Η ταυτότητα των γυναικών Ρωμά είναι μια σύνθετη ταυτότητα και διακλαδική, όπου περιλαμβάνονται πολλές μορφές διάκρισης και κυριαρχίας, ο ρατσισμός, ο σεξισμός και έχουν συγκεκριμένες ε, ταυτότητες. Πολλές γυναίκες έχουν τέτοια επίγνωση. Μία από αυτές μας έλεγαν ότι το να είναι σήμερα γυναίκα κάποια ε, Ρωμά είναι καθημερινή μάχη. Γιατί είναι περίπλοκο, σύνθετο να είσαι και Ρωμά και γυναίκα. Ταυτόχρονα ωστόσο είναι και περηφάνεια. Γιατί για μένα το να, είναι, το να είμαι γυναίκα και να είμαι ε, Ρωμά είναι τιμή, είναι προνόμιο. Μια, ένας άλλος κεντρικός άξονας στη διαμόρφωση αυτή τη σύνθετη ταυτότητα είναι η οικογένεια. Όχι ως πυρηνική οικογένεια όπως ε, θεωρούμε, αλλά σε, η ευρεία εκτεταμένη οικογένεια, η οικογένεια ο θεσμό οικογένεια στην κοινότητα των Ρωμά δεν αποτελεί μόνο το κέντρο διοργάνωση καθημερινή ζωή, αλλά και τον βασικό κοινωνικοποιητικό παράγοντα και παράγοντα συσχετισμού των μελών τη και κοινωνική αναγνώριση. Η οικογένεια είναι ο χώρος στον οποίο διαμορφώνονται οι ταυτότητες και ορίζονται οι προσδοκίες αλλά και οι μορφές συμπεριφορά ανδρών γυναικών. Συνιστούν ταυτόχρονα ένα πλαίσιο, ένα χώρο προστασίας και αλληλεγγύης σίγουρα και ένα χώρο κοινωνικού ελέγχου που μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της αυτονομίας και τις ελευθερίας των γυναικών Ρωμά. Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε και πρέπει να αναλύσουμε καταστάσεις βίας που βιώνουν οι γυναίκες Ρωμά. Όπως ήδη ανέφερα σε ένα από τα πρώτα θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να αναλύσουμε την, ε, ε τη διαφορετικότητα της εμπειρίας βίας κατά των γυναικών είναι οι θέσεις της κοινο, των κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών. Δηλαδή, το να ξέρουμε πώς η κοινότητα, η συγκεκριμένη κοινότητα, η κοινότητα των Ρωμά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ορίζει, καθορίζει, κατανοεί και τοποθετείται σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών. Αυτό μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για το βαθμό νομιμοποίησης της βίας και ιδίως για τις δυνα... πραγματικές δυνατότητες των γυναικών Ρωμά να αντιμετωπίσουν τη βία. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε το πρόγραμμα Δάφνη που σας περιέγραφα, είδαμε διαφορετική συμπεριφορά των γυναικών, της κοινότητας μας στη βία των γυναικών. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι αυτό που λέμε δεν είναι ούτε εξαντλητικός ούτε αποκλειστικός κατάλογος. Πιστεύουμε ωστόσο ότι περιλαμβάνει τις πιο σύνηθεις, ε, τις πιο συνήθεις συμπεριφορέ ε, συμπεριφορές των Ρωμά στη βία. Διευκρινίζουμε ότι δεν είναι μια αναλυτική εικόνα. Οι αντιδράσεις παρουσιάζονται ε, συν, ε, συνενούμε, συνενούμενες. Ταυτόχρονα δεν είναι αποκλειστικές αντιδράσεις της κοινότητας των Ρωμά, αλλά μπορούν να αναγνωριστούν περισσότερο ή λιγότερο και από την πλειοψηφούσα, από το πλειοψηφούν της κοινωνίας σας. Μίλησε για την νομιμοποίηση της βίας, για την τυποποίηση της βίας. Είναι κάτι κατανοητό και σχεδόν συγνωστό. Του αόρατου χαρακτήρα της βίας συχνά υπάρχει σιωπή γύρω από το φαινόμενο της βίας. Δεν, είναι, δεν μιλάμε για το φαινόμενο και άρα δεν υπάρχει η ευθύνη, η ανάληψη ευθύνη των γυναικών ενώπιον της βίας και η άρνηση, η αμή αποδοχή της βίας. Ως συνέπεια της απομόνωσης και του κλίματος ε, ε, τυποποίησης, δύσκολα μπορεί μια γυναίκα να βγει από την κατάσταση βίας που βιώνει. Το να καταφέρει η γυναίκα Ρωμά να καταλάβει και να αποδεχθεί ότι υφίσταται μία ανδρική βία είναι μία μακρά δύσκολη διαδικασία που έχει πολλά εμπόδια διάφορων ειδών. Πρώτον, πρέπει να τονίσουμε ότι η ιστορική διαδικασία δίωξης και περιθωριοποίησης του λαού των Ρωμά δημιούργησε μια συλλογική ταυτότητα αντίστασης που υλοποιείται στην ε, ανάπτυξη στρατηγικών επιβίωσης και διαφύλαξης της κουλτούρας μέσα στην, στο εσωτερικό της πλειοψηφούσας κουλτούρας, της κουλτούρας της πλειοψηφίας. Οι στρατηγικές επιβίωσης και αντίστασης μπορεί να είναι χρήσιμες. Είναι χρήσιμες για να διαφυλάξουν την ταυτότητα, την πολιτιστική ταυτότητα των Ρωμά, αλλά δεν είναι ουδέτερες ό,τι αφορά το φύλλο. Επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο άνδρες και γυναίκες Ρωμά και έχουν αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο όπως είδαμε, στις γυναίκες και την αυτονομία τους. Πρόκειται για στρατηγικές που μετατρέπονται στην οικογενειακή πίεση να διατηρηθεί το status που επιτρέπει την αναπαραγωγή της πατριαρχικής τάξης όπως διαμορφώνεται στις κοινότητες των Ρωμά και σε πίεση για την επίλυση των συγκρούσεων βίας από την υπεροχή της κυριολογικής ταυτότητας και του συμφέροντος της ομάδας και όχι τον, εις των ατομικών δικαιωμάτων των γυναικών που συγκρούνται με την αρχή αυτή. Αυτές οι πολιτιστικές στρατηγικές δεν είναι ουδέτερες όπως είπα, έχουν μεγάλο αντίκτυπο και σημαντικό βαθμό ε, επιρροή στην κατανόηση, την επίγνωση και την αποδοχή της πρόσβασης σε συγκεκριμένα δικαιώματα που έχει μια γυναίκα στην κοινωνία στην οποία μετέχει η κοινότητα Ρωμά. Πρόσβαση που που δυσχεραίνεται περισσότερο από το ρατσισμό που υφίσταται ο λαός των Ρωμά και που εκδηλώνεται και στις υπηρεσίες πρόσβασης, μέρημνας κλπ. Αυτό εξηγεί την έλλειψη εμπιστοσύνης των γυναικών Ρωμά προς τις δημόσιες υπηρεσίες εν γέννη και την ε, άρνηση λόγω των δυσκολιών στην καταγγελία της βίας που δεν θεωρείται ως μία δυνατότητα ουσιαστικής προσφυγής, αλλά μία στιγματοποίηση της γυναίκας. Επίσης, να τονίσουμε ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες προστασίας των θυμάτων ανδρικής βίας, οι υπηρεσίες που προέρχονται από την πλειοψηφική κοινωνία, δεν είναι έτοιμες για να, δεν είναι προετοιμασμένε για να καλύψουν, να δώσουν απάντηση στα αιτήματα των γυναικών Ρωμά και στα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Εμείς θεωρούμε ότι η προοπτική αυτή δεν, ότι οι γυναίκε Ρωμά ε, θεωρούν πως δεν υπάρχει επαρκής προστασία και επαρκής αντιμετώπιση από τις υπαλλήλου τους οποίους ε, προσέφυγαν. Κλείνω με κάποιες γραμμές, ε, με κάποιες θέσεις πιθανής μελλοντική δραστηριότητα που προέκυψαν σαφώς ως αποτέλεσμα της ε, επιτόπιας δουλειά που κάναμε και κατά την άποψή μας είναι ουσιώδους χαρακτήρα για να προχωρήσουν και στην υπέρβαση της βίας κατά των γυναικών, όσο και για τη διαδικασία ένταξης των ε, γυναικών Ρωμά. Πρώτον, κατά την άποψή μας πρέπει να διευκολυνθούν περιβάλλονται εμπιστοσύνη, όπου οι γυναίκες μαθήματα της ε, ανδρικής βίας θα μπορούν να αισθανθούν άνετα, να αισθανθούν ότι αναγνωρίζονται, ότι γίνονται κατανοητές και αποδεκτές από τις κοινωνίες, σαν πρώτο βήμα για να μπορέσουν να εκφράσουν την εμπειρία της βίας. Αν αυτό το περιβάλλον, το θετικό περιβάλλον δεν υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο οι γυναίκες Ρωμά να αποφασίσουν να εκφράσουν αυτή την κατάσταση βίας. Επίσης, πρέπει να δουλέψουμε σε προγρά... ειδικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για να διαλυθούν, για να, για να υπονομευθούν οι στρατηγικές νομιμοποίησεις ε, και επαναθυματοποίησης που, που διονίζουν τη βία κατά των γυναικών. Επίσης, ο στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργηθούν δράσεις προς γυναίκες που οργανώνονται και διαμορφώνονται από στρατηγικές ενίσχυσης της ατομικής ε, ε, δύναμής τους, με αύξηση της στρατηγικής ενίσχυσης, της ταυτότητάς τους, των δυνατοτήτων τους, των στοιχείων που έχουν ως μηχανισμό ε, εξόδου από το αδιέξοδο. Είναι κλειδιά αυτά για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην αναγνώριση της δικής τους ατομικής ταυτότητας ως γυναίκα Ρωμά. Μια άλλη βασική γραμμή είναι η ειδική παρέμβαση ανδρών Ρωμά με την ευαισθητοποίηση που τους ανοίγει δρόμους για να επανεξετάσουν την ε, δική τους ανδρική ταυτότητα μέσα στην ίδια κοινότητα των Ρωμά. Κάτι απαραίτητο, κατά την άποψή μας. Και μια τελευταία παρατήρηση. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε, να δουλέψουμε στην ανάπτυξη της, ε, των διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εργαζομένων στο χώρο της ε, προστασίας των γυναικών τους ώστε να προσαρμόσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες όπως ε, τις δομές υποδοχής ή τα κέντρα προστασίας γυναικών και να μην αισθάνονται, ούτως ώστε να μην αισθάνονται οι γυναίκες Ρωμά αόρατες στο πλαίσιο αυτό. Αυτή τη στιγμή πολύ λίγες γυναίκες Ρωμά υπάρχουν που έχουν πρόσβαση, πηγαίνουν σε αυτές τις υπηρεσίες, πηγαίνουν στις, στα επίγοντα, στις, στις γραμμές, ε, ε, στα τηλέφωνα επίγουσας ανάγκης ή στους, χώρες, ε, στους χώρους υποδοχής γυναικών θυμάτων βίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Όταν πριν από λίγο, λίγα χρόνια είχαμε αναλάβει την έκθεση για τους Ρωμά, είχα έναν συνάδελφο φιλελεύθερο, ευρωβουλευτή, που συνεργάστηκε μαζί μας και ε, τότε είχαμε συμπεριλάβει τις πατριαρχικές παραδόσεις στην έκθεση και την είχε καταψηφίσει την έκθεση, διότι θεωρούσε πως... Ε, η κατάσταση αυτή που περιγράφαμε εμείς δεν ήταν αντιπροσωπευτική. Όμως, όλοι γνωρίζουμε πώς η έμφυλη διάσταση είναι υποτιμημένη. Και για αυτό πιστεύω πως ε, είναι και ο λόγος που έχει αποτύχει η στρατηγική. Επίσης υπάρχει έλλειψη σύνδεσης ε, της ε, πολιτικής με την πράξη, με τους ανθρώπους αυτούς και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολύ περισσότερα μαθαίνουμε από τους αυτόπτες μάρτυρες βλέποντας ε, τι γίνεται από ότι τα προηγούμενα χρόνια όπου είχαμε μεγαλεπίβολα σχέδια και μία προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω όπου στην ουσία δεν βλέπαμε τους ε, Ρωμά, δεν βλέπαμε τι γίνεται, δεν βλέπαμε την αλήθεια και την πραγματικότητα και δεν μπορούσαμε επομένως και να την αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, αναφέρθηκα πριν στην ε, καθημερινή βάση λήψη των εκθέσεων και χρειάζεται αυτό, χρειάζεται αυτή η καθημερινή λήψη εκθέσεων, αντικειμενικών εκθέσεων έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη αξιολόγηση. Υπήρχαν στο παρελθόν οργανώσεις και υπηρεσίες που συνέτασαν εκθέσεις για τους Ρώμα χωρί να έχουν δει ποτέ κανέναν, χωρίς να έχουν πάει ποτέ εκεί. Τώρα όμως ε, με μεγάλη μου χαρά σα λέω ότι έχουμε επί τόπου που βρίσκονται εκεί και ξέρουν τι λένε. Και είναι κάτι που πραγματικά είναι πολύ ανακουφιστικό. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ γι' αυτό. Η επόμενη ομιλία τώρα θα είναι αφιερωμένη στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία έχουν αποφασίσει να εργαστούν μαζί μου και να συνεργαστούμε για αυτό το θέμα και να συνεισφέρουν άτομα που είτε συμμετείχαν και στην προηγούμενη έκθεση ως κοιόδης εισηγητές και άτομα που συνεργάζονται μαζί μας τώρα. Είχαμε την πρώτη συνάντηση σκιωδών εισηγητών σήμερα το απόγευμα. Η Κορνέλια Ένστη είναι εδώ η Ρενάτε Βέμπερ επίσης ε, συμμετέχει στην ομάδα και θα τους δώσω το λόγο τώρα να μας μιλήσουν. Αν θέλεις Κορνίλια, έχεις το λόγο ή όπως θέλετε, όποιος θέλει. Ραούλ, άρχισε πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όχι μόνο για τη διοργάνωση της ε, συνεδρίασης αυτής, αλλά και για τα θέματα που έχετε επιλέξει. Όντως, εδώ και πολλά χρόνια συζητάμε το θέμα αυτό και το πρόβλημα δεν είναι κατά ανάγκη έλλειψη προτάσεων και ιδεών. Το πρόβλημα βασικά είναι η έλλειψη πολιτικής εθέλησης για να εφαρμοστούν αυτές οι ιδέες και αυτές οι προτάσεις. Και αυτό η αλήθεια είναι, είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο, Ορισμένες ε, πτυχές ε, πρέπει να αναφερθούν, οι πολιτικές είναι κάποιες από αυτές τις πτυχές και κάποιες άλλες είναι πιο τεχνικές. Πιστεύω όμως, όπως και να έχει, πως όλες είναι εξίσου σημαντικές. Όσον αφορά τώρα την αντίληψη ε, του θέματος, δεν είναι, θα το έλεγα κάποιος, δεν θα το έλεγα εθνικό πρόβλημα, είναι κάποια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, Χαρήκα πολύ που άκουσα αυτές τις ε, δύο ομιλίες. Μία της ε, συναδέλφου που είναι και αυτή από την Βαρκελόνη, της κυρία Σουρία και χάρηκα πολύ όχι μόνο επειδή ξέρω πολύ καλά τη δουλειά που, γίνε, που κάνουν εκεί, αλλά ξέρω επίσης και τα αποτελέσματα που έχει η δουλειά τους και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα γίνεται στη δουλειά τους. Τώρα υπάρχουν ορισμένοι βασικοί τομείς που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και με τη Λίβια, οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι βασικοί άξονες τη συζήτησή μας. Ε, καταρχάς το ζήτημα της ε, διάκρισης όσο πυρήνας, η ρίζα του προβλήματος το πρόβλημα δεν είναι μόνο η πρόσβαση ε, στις υπηρεσίες ε, υγείας, στην ιατρική περίθαλψη. Πολλές φορές βλέπουμε και έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα, έλλειψη εμπιστοσύνη στο ότι, στην πρόσβαση στο σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές επιτυχίες με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Το πλαίσιο όμως πολλές φορές οφείλεται, ε, έχει να κάνει με πραγματικές ε, περιπτώσεις διακρίσεων. Και ας ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες Ρωμά αυτές που πλήττονται από διακρίσεις. Αυτές περισσότερο επειδή είναι όχι μόνο γυναίκες αλλά και Ρωμά. Έπειτα, να μην ξεχάσουμε το ζήτημα της φτώχειας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις ε, διακρίσεις. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί επίσης σε συνδυασμό με τις διακρίσεις. Ε, σωστά είπατε πως δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τους λόγους για τους οποίους γίνονται διακρίσεις. Αντίθετα, πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε τι γίνεται με την αρχή των πολλαπλών διακρίσεων. Είναι κάπως περίπλοκο νομικά το θέμα, ωστόσο πρέπει να αναλυθεί. Υπάρχει νομική κάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως η εξωτερική διάσταση είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Η πραγματικότητα είναι απόλυτα διαφορετική και αυτό για μένα είναι ένα από τα κεντρικά σημεία, είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να αναλύσουμε. Επίσης, κάτι άλλο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι το εξής. Όσον αφορά το ρόλο των ε, οργανώσεων, των οργανισμών αυτών, να πω ότι πολλές φορές ε, γκρινιάζαμε για την έλλειψη συμμετοχής από οργανώσεις ε, Ρωμά που θα βοηθούσαν στον ορισμό, στον εντοπισμό ε, του προβλήματος, στον, ορισμό, στον καθορισμό στρατηγικών και στην εφαρμογή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι το να δώσουμε περισσότερη δύναμη περισσότερη χειραφέτη σε αυτούς τους ε, οργανισμούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές το πρόβλημα είναι η έλλειψη αξιοπιστίας και η έλλειψη αξιοπιστίας οδηγεί και σε ελλειπή εφαρμογή των ε, στρατηγικών. Τώρα το τρίτο σημαντικό ζήτημα είναι κάτι το οποίο μαστίζει ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου, η ανάγκη χρηματοδότησης. Πολύ συχνά έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με έλλειψη χρηματοδότησης και τουλάχιστον στη δική μου περιοχή αυτό που βλέπουμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ καλά προγράμματα και καλές στρατηγικές, η έλλειψη πόρων είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και επηρεάζει άμεσα την εφαρμογή τους και αυτό πολλαπλασιάζει γεωμετρικά τα, τις αρνητικές επιπτώσεις. Τα κονδύλια λοιπόν. τα οποία δεν είναι μόνο ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών, είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε και να παραβλέπουμε σε καμία περίπτωση. Τέλος, πιστεύω πως είναι εξίσου σημαντικό και δεν θα ίσω τα λόγια μου σε αυτό το σημείο, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο ότι υπάρχει συγκεκριμένη και στοχευμένη βία στις γυναίκες ανάλογα με τις συνθήκες ζωής τους. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι η ατιμορρησία. Η ατιμορρησία είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και απόλυτα. Όχι μόνο με, όχι μόνο με την αστυνομία, αλλά και από την κοινωνία την ίδια. Πρέπει να αντιμετωπιστεί δηλαδή όχι μόνο σε επίπεδο αρχών, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Πρέπει να αλλάξουν η ρόλη να αλλάξει αυτό το πατριαρχικό σύστημα το οποίο έχει οδηγήσει και σε αυτή την ατιμορρησία. Αυτά είναι κάποια βασικά θέματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν συζητάμε το όλο ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Είστε ένας από τους ευρωβουλευτές που ασχολείται με το θέμα αυτό εδώ και εννιά χρόνια. Γνωρίζετε λοιπόν για τι πράγμα μιλάτε. και το πώς έχουν τα πράγματα στην Ισπανία. Και η Κορνέλια είναι εμπειρογνώμων που έχει συμβάλει σημαντικά στο ίδιο το πλαίσιο όταν το ετοιμάζαμε στην Επιτροπή πριν δύο χρόνια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Λίβια και Κίνγκα. Χαίρομαι που συζητάμε σήμερα εδώ αυτό το θέμα. Χάρηκα με τις ε, παρεμβάσεις της κυρίας Κόσμα και της ε, κυρίας Σεράνο. Ήταν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ε, στο θέμα αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω από την παρέμβαση της κυρίας Κόσμα. Αναφέρατε την σχολική εκπαίδευση ως πολύ σημαντικό στοιχείο. Συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι στοιχείο κλειδί σε όλες τις χώρες και χαίρομαι που πράγματι κάτι συμβαίνει στον τομέα αυτών. σε κάποιες χώρες, σε άλλες χώρες μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Όπου αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι οι Ρωμά ε, πρέπει να πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία. Αυτό συνεχίζει να ισχύει στην ε, Τσεχία, χώρα γειτονική με τη δική μου. Και έτσι ε, δεν λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση. Πώς ε, λοιπόν είναι τα πράγματα ε, σε εσάς, ε, στη χώρα σας, πώς ήταν, τι εμπειρίες έχετε συλλέξει. Κάποιοι λαμβάνουν καλή εκπαίδευση, αλλά στην αγορά εργασίας νέες γυναίκες δεν βρίσκουν εργασία. Νομίζω ότι ο ρατσισμός παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι κάτι που πάντα ε, επικρίναμε στην ε, στρατηγική των Ρωμά. Η καταπολέμηση του ρατσισμού θα πρέπει πάντα να είναι σημαντικό στοιχείο στα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να ρωτήσω πρακτικά τι μπορεί να κάνει κανείς για να καταπολεμήσει το ρατσισμό οι γυναίκες Ρωμά ε, δέχονται διπλές διακρίσεις και λόγω του φίλου τους. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω τι γίνεται με την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες είναι ε, πολύ κακή η κατάσταση, για να το πω και ήπια. Ε, εσείς ε, τι εμπειρίες ε, έχετε συγκεντρώσει στο θέμα αυτό και κύριε Σεράνο. Σωστά είναι όλα αυτά που μας περιγράψατε, η ειδική θέση των γυναικών Ρωμά. έχω κάνει πολλά ταξίδια και παρόμοια πράγματα έχω δει και εγώ. Αλλά για τις γυναίκες Ρωμά μπορούμε να διευκολύνουμε τα πράγματα αν γνωρίζουν ότι είμαστε αδελφές και ότι πριν μια-δυο γενιές είχαμε και εμείς τα ίδια προβλήματα. Ε, και από τη δική μας ιστορία ε, γνωρίζουμε τέτοιες συνθήκες. Ε, ίσως λοιπόν θα έπρεπε να εργαστούμε με αυτό το κοινό σημείο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τις γυναίκες αυτές. Ήθελα να το τονίσω αυτό. Ε, και ε, θα πρέπει να δούμε τι, τι κοινά προβλήματα έχουμε να καταπολεμήσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω τις ε, διαφορές μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου. Μικρόφωνο παρακαλώ. I'm very sorry. I, didn't know that you did. Ζήτω συγγνώμη. Ε, σας έδωσα λοιπόν το λόγο και εσείς ε, ασχολείστε με το θέμα αυτό εδώ και πολλά ε, χρόνια και ε, οι παρατηρήσεις σας ε, πάντα κινούν τη συζήτηση. Εσείς λέτε πάντα και πού βρίσκονται οι Ρώμα, τι κάνουν, αλλά η, όλο όλη αυτή η στρατηγική έχει ξεκινήσει από τους ίδιους του Ρωμά. Και πιστεύουμε ότι η οικιακή βία, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ε, κλπ. Ε, οφείλεται σε εκατοντάδες χρόνια στο περιθώριο της κοινωνίας. Εάν κοιτάξετε την ιστορία της Ουγγαρίας, για παράδειγμα, την ιστορία της Σλοβακίας, ε, την ιστορία της Δυτικής Ευρώπης, θα δείτε ότι η Ρωμά ε, ήταν παρόντες επί 800 χρόνια. Συμμετείχαν το 1956 στη, στο δημοκρατικό αγώνα στην ε, Ουγγαρία, ε, το 89 στην Τρανσιλβανία. Ε, οικοδόμησαν και αυτοί τις χώρες στα εργοστάσια τη δεκαετία του 70, του 80, στην Ανατολική Ευρώπη. Ε, άλλωστε ε, υπό το κομμουνιστικό καθεστώς έπρεπε να εργαστεί κανείς, αλλιώς πήγαινε φυλακή. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν για μένα τώρα να βλέπω πώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μπορούν να παρουσιάσουν αυτή την ιστορία 800 ετών. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, διότι κάθε φορά που παίρνετε το λόγο ε, λέτε πράγματα τα οποία ε, δίνουν ε, ορμή στη συζήτηση. Άλλωστε στο Κοινοβούλιο ε, άλλωστε στο Κοινοβούλιο ε, εξαρτώμαστε από τη συνεργασία 6-7 πολιτικών ε, ομάδων. Ζητώ συγγνώμη που τα είπα αυτά ως πρόεδρος, είμαι η συγγήτρια του θέματος, ως η συγγήτρια τα λέω. Μια πολύ σύντομη ερώτηση και μία που είναι ίσως δύσκολο να τεθεί. Ακούσαμε από την κυρία Ρούμπιο Σεράνο όχι μόνο τα περί οικιακής βίας, αλλά και τον τρόπο που ε, ε, έδινε μεγάλη αξία στην ε, εγκράτεια από πλευρά των γυναικών. Στην Παρθενιά. Έπρεπε να ακολουθούν τους κανόνες αυτούς. δεν το αμφισβητώ, αλλά δυσκολεύομαι να το συνδυάσω με το γεγονός ότι γίνεται εμπορία γυναικών Ρωμά. Εάν λοιπόν οι άντρες Ρωμά εκπροσωπούνται δυσανάλογα πολύ ε, μεταξύ των ε, εμπόρων ανθρώπων ε, και οι γυναίκες εκπροσωπούνται δυσανάλογα μεταξύ των θυμάτων, ποια είναι η σχέση μεταξύ των εμπόρων ανθρώπων και των θυμάτων. Ανήκουν σε κάποια υπομάδα, κάποια ομάδα με χαμηλότερη θέση στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν έθεσα σαφώ την ερώτηση. Ε, στο πλαίσιο αυτό ρωτώ, αν, μιλούσαμε για τους ε, Αλβανούς ε, θα ρωτούσα για αυτούς, αλλά τώρα μιλάμε για τους Ρωμά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, είμαι ε, βέβαιη ότι οι ε, εμπειρογνώμονες μας θα μπορέσουν να απαντήσουν. Η Πλάνκα ξέρω ότι εργάζεται ως δικηγόρος, ως νομικός και θα μπορέσει να απαντήσει, αλλά επιτρέψτε μου να ρωτήσω, θέλετε να απαντήσετε ή να ακούσετε όλες τις ερωτήσεις πρώτα. Ωραία, να δώσω το λόγο πρώτα στις δύο κυρίες να απαντήσουν. Ε, προτού να ακούσουμε τα περί της νέας έκθεσης ε, τη ΕΦΡΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Πήραμε πολλές ερωτήσεις χρήσιμες. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δεν μπορούσα να, συμπληρω... να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου γιατί είχα πάρα πολλά πράγματα να πω. Ήθελα να μιλήσω για τη βία την εκπόρνευση γυναικών. Μιλάμε για χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις εντός και εκτός Ουγγαρίας. Έχουμε μια, ιστορία, μια παροιμία στην ε, Ουγγαρία που λέει το ένα μου μάτι κλαίει, το άλλο γελάει. Εμένα και τα δύο μάτια κλαίνε όταν βλέπω την ε, αντιμετώπιση παιδιών και γυναικών. Στην πραγματικότητα στην Ουγγαρία οι γυναίκες Ρωμά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και με δύο και με τρεις δουλειές ακόμα. Ούτε μπορούν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα μόνες τους. Οπότε, ο μόνος τρόπος για να πετύχουν κάτι τέτοιο είναι η πορνεία. Και αυτό όμως είναι κομμάτι της βίας. Τώρα για τη χρήση των πόρων της Ένωσης, έχουμε πολύ αρνητική εμπειρία. Τα χωριά δεν παίρνουν σχεδόν τίποτα. Στις μεγάλες πόλεις, στη Βουδαπέστη, Έρχονται δισεκατομμύρια, αλλά πολλές φορές αυτά τα δισεκατομμύρια χρησιμοποιούνται εις βάρος των Ρωμά. Ε, στις πόλεις που υπάρχουν λεφτά, σχολεία, δουλειές, διώχνονται οι Ρωμά σιγά σιγά. Διότι όταν λέμε αποκατάσταση μιας περιοχής, σημαίνει ότι ο Ρωμά που μένει εκεί διώχνεται με τον ΑΒ τρόπο από τη συγκεκριμένη γειτονιά. Έμενα στο κέντρο της Βουδαπέστης ήμουνα και δημοτική σύμβουλος. Πήραμε πάρα πολλά χρήματα για την αποκατάσταση κτηρίων του κέντρου της πόλης. Ούτε μια δουλειά στα έργα αυτά δεν μπόρεσα να βρω να το κάνει ένας Ρωμά. Έχουμε λοιπόν μεγάλα έργα που δεν εμπλέκουν Ρωμά. Προσπάθησα να αναφέρω πόρους των Ρωμά σε ΜΚΟ. Οι μικρές ΜΚΟ δεν έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους. Οι μεγάλες ΜΚΟ που δεν έχουν Ρωμά όμως έχουν πρόσβαση σε τέτοιους ε, πόρους. Δεν λέω ότι οι μεγάλες ΜΚΟ δεν χρησιμεύουν για τους Ρωμά, αλλά δεν έχουν Ρωμά, δεν έχουν εικόνα της κατάστασης, δεν συνεργάζονται μαζί μας και πολύ λίγοι διανοητές Ρωμά μπαίνουν ή τέλο πάντων ε, μελετητές Ρωμά μπαίνουν σε αυτές τις μεγάλες ΜΚΟ και τελικά τα κονδύλια της Ένωσης θα έπρεπε να περιλαμβάνουν και κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχουν δικαιούχους όχι μόνο ΜΚΟ που δουλεύουν για τους Ρωμά, αλλά και με Ρωμά. Τώρα, δεν σας πω την ιστορία της ζωής μου, αλλά είχα δουλέψει σαν καθηγήτρια σε σχολείο. Και μπορώ να σας πω ότι αν ένα παιδί, ένα παιδί σε μια τάξη που δεν εντάσσεται, φεύγει από την κοινότητα της τάξης. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν σχολεία με, ρομπά, με Ρωμά όπου όμως τα παιδιά είναι τελείως απομονωμένα. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Έχουμε άλλες περιπτώσεις όπου Ρωμά διώχνονται από τις πόλεις σε άθλια χωριά γιατί, γιατί εκεί υπάρχουν σχολεία με αρκετά παιδιά Ρωμά και άρα τους βάζουμε και τους άλλους εκεί μαζί. Εάν δεν υπάρχει ένταξη εξ αρχής υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάθε παιδί πρέπει να μπορέσει να έχει ένα δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να μπορέσει να περάσει, να υλοποιηθεί η, η, η ένταξή του. Σας είπα ότι πολλά πράγματα είχα να πω, πάρα πολλά πράγματα είχα να πω. Θα μπορούσα να μιλήσω για τα συστήματα κοινωνικής ε, για τα, τα συστήματα κοινωνικής ε, ανέλυξης. Υπάρχουν πολλά ελιτίστικα σχολεία στο, στην ε, Ουγγαρία που χρηματοδοτούνται από, ε, από το κράτος. Εκεί δεν μπορούν να μπουν παιδιά Ρωμά. Ακόμα και αν είναι έξυπνα. Ένα παιδί δωμά που θέλει να γραφτεί εκεί του λένε δεν έχουμε θέσεις, πηγαίνετε αλλού. Όσο δεν υπάρχει υποχρέωση τέτοια σχολεία να δέχονται όλα τα παιδιά εφόσον χρηματοδοτούνται από το δημόσιο κορβανά, έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Ε, Πιστεύω ότι θα έπρεπε, δεν θέλω να κατακρίνω τα μεγάλα, τις μεγάλες ΜΚΟ, πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε σοβαρές αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε πόδους. Τώρα, για τους πόρους της Ένωσης. Στις εθνικές στρατηγικές δεν βρήκαμε τις προϋποθέσεις να υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν την αρχή της ισότητας των φύλων όταν θέλουν να πάρουν ευρωπαϊκούς πόρους. Ελπίζω αυτό να το πετύχουμε. Στην Ουγγαρία Το πετύχαμε αυτό. Από τον Ιούλιο και μετά καμία πόλη δεν μπορεί, της Ουγγαρίας δεν μπορεί να πάρει χρηματοδότηση ενωσιακή αν δεν έχει ε, πολιτική, ε, πολιτική ε, ισότητα των φίλων. Εγώ ξέρετε είμαι και ειδική για θέματα ισότητας Οι πόλεις είναι αυτές που διαμορφώνουν τις πολιτικές ισότητας ευκαιριών και αυτές αποφασίζουν πώς θα κατανείμουν τους πόρους για να καλύψουν τον όρο ισότητα. Ρωμά, άτομα με αναπηρίες κλπ. Ανέφερα ήδη ότι υπάρχουν τα προγράμματα αποκατάστασης των πόλεων τα προγράμματα αυτά διαμορφώνονται από τις δημοτικές αρχές. Δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης σε τέτοια. Διαφωνούμε με την αρχή αυτή. Θέλουμε οι Ρωμά να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά. Δεν είμαστε όμως αρκετοί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυστηρούς κανόνες από εσά, από το δικό σας επίπεδο χρειάζεται να ξέρουμε τι αναμένει η Ένωση για να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια των ε, Ρωμά. Αυτή τη στιγμή προτείνουμε ένα πίνακα ένταξη των Ρωμά, το dashboard που λέμε, στην Επιτροπή, που είναι πολύ σημαντικό γιατί μερικέ φορέ βλέπουμε να χρησιμοποιούνται προγράμματα της Ένωσης εις βάρος των ε, Ρωμά. η κυρία Σεράνο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Πρώτον, τέθηκε ένα θέμα για το πώς θα χτυπήσουμε το ρατσισμό, ιδίως στο χώρο της εργασίας. να σας πω μια εμπειρία που θεωρούμε ενδιαφέρουσα. Από το 97 έγινε μέσω ενός από τα πρώτα ευρωπαϊκά έργα του Λεωνάρντο με νέες γυναίκες Ρωμά. Χιτάνας Αμπριέντο Καμίνο το ονομάσαμε. Και ξεκινούσαμε από αυτή την διάσταση αντιμετώπιση του ρατσισμού. Προσπαθούσαμε να περάσουμε επαγγελματικά προσόντα σε γυναίκες Ρωμά. Οι ίδιε αποφάσισαν τι θέλαν να κάνουν. Είπαμε, ωραία, θα κάνουμε ό,τι θέλετε. Είπαμε, θα κάνουμε ό,τι θέλετε, αλλά καλά. Ετοιμάσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα κατάρτιση με ένα από τα καλύτερα κομμωτήρια τη Βαρκελόνη και της Ισπανίας, του Αλονγκέρος, για να μπορέσουμε να πούμε μετά, ναι, είναι Ρωμά, αλλά είναι και καλύτερες επαγγελματίες. Αυτό το θετικό μήνυμα ε, τους άνοιξε το δρόμο στο χώρο εργασίας. Αυτή η θετική εικόνα, η ανάδειξη της συνεργασίας με κάποια άτομα για να αναδείξουν με τη σειρά τους την αξία των γυναικών Ρωμά μας βοήθησε πάρα πάρα πολύ για να χτυπήσουμε τη διάκριση. Κάτι άλλο η προσοχή στο μεταξύ του κοινού και του διαφορετικού. Ε, όντως οι γυναίκες έχουν πολλά κοινά, αλλά ταυτόχρονα είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση και στο διαφορετικό. Γιατί οι, οι γυναίκες Ρωμά, το είπαμε, πρέπει να μπορούν να κάνουν το δικό τους, να πάρουν το δικό τους δρόμο. Όπως ακριβώς η πατριαρχική οικογένεια μπαίνει στην κοινωνική και ατομική ζωή, οι ίδιες οι γυναίκες Ρωμά είναι αυτές που πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, λέγοντας πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και ως γυναίκες και ως ε, Ρωμά. Για να μπορέσει να φύγει η βία, να εξαφανιστεί η ε, διάκριση. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο για τις ε, γυναίκες. Τρίτο θέμα που θέλω να θέσω και που εμφανιζόταν στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων και της ε, ε παρθενίας. Να σας πω ότι στην Καταλωνία τουλάχιστον δεν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες Ρωμά στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Βέβαια, είναι περίπλοκο το θέμα της εμπορίας. Πάντως σας λέω, δεν υπάρχει υπερεκπροσώπηση των Ρωμά εκεί. Οι γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας είναι κυρίως γυναίκες από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και Ευρωπαίες. Αλλά στην Καταλωνία δεν υπάρχει αυξημένος αριθμός γυναικών Ρωμά. Εμεί μιλάμε για μια κοινότητα Ρωμά που υπάρχει στην Ισπανία τουλάχιστον 600 χρόνια και, άρα είναι μια κοινωνία που βρίσκεται εκεί, στην Ισπανική κοινότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα για το θέμα της Παρθενίας. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά. Δεν είναι παράξενο. Συμβαίνει στις δυτικές κοινωνίες πάντα συνέβαινε. Στη δυτική κοινωνία οι άνδρες, επειδή ακριβώς θεωρούν ότι η γυναίκα είναι κτήμα τους, ελέγχουν την ε, σεξουαλικότητά τους. Και η εκπόλευση είναι κομμάτι αυτού του ελέγχου. Αυτή είναι η κατάσταση που καταγγέλουμε. Και αυτό συμβαίνει. Υπάρχει αυτή η κατάσταση γιατί υπάρχει η πατριαρχική κοινωνία και δεν είναι μόνο στου ε, Ρωμά. Περισσότερο ίσω, αλλά αυτό συμβαίνει και σε υπόλοιπε και σε άλλε δυτικέ κοινωνίε. Αυτό σημαίνει έλεγχο στι γυναίκε, Αλλά αυτό συμβαίνει και στι δυτικέ κοινωνίε που είναι πατριαρχικέ. Δεν είναι παράξενο το ότι αυτό συμβαίνει και στου Ρωμά. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το άφησμα αξιών διαμορφώνει μια διαφορετική πραγματικότητα. Δεν είναι όμω κάτι ξένο, είναι σύνηθε. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία να τα λέμε όλα αυτά. Νομίζω ότι οι περισσότερες προκαταλήψεις ε, προέρχονται από την έλλειψη γνώσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ε, ε, ακούμε νέα πράγματα και θα προχωρήσουμε πιο βαθιά τώρα. Έχουμε τη νέα μελέτη του FRA Είναι ίσως η μόνη μελέτη που έχει τα τελευταία δέκα χρόνια που να αξίζει τα λεφτά της. Και το λέω προς τα τμήμα πολιτικής ότι ήδη έχουμε εκπονήσει κάποιες εκθέσεις που δεν νομίζω ότι ήταν καλή ιδέα. Ε, δεν ε, μάθαμε πολλά στοιχεία από αυτές. Στις, και στις δύο άλλες εκθέσεις του Ρωμά που είχαμε, είδαμε επικάλυψη εργασιών, είδαμε ότι διάφοροι οργανισμοί κάναν την ίδια δουλειά και την δημοσίευσαν εκατοντάδες φορές. Ε, τούτη τη φορά όμως έχουμε νέες γνώσεις για επίμαχα ζητήματα και μερικές φορές είναι επίμαχα και τα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Δημητρακόπουλο. που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα των Ρωμά όπως και η Λίνα. Να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για τη δουλειά σας, ε, σας ευχαριστούμε γενικά για όλη τη δουλειά που κάνετε για την ε, ισότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας δίνω το λόγο και με την έκθεσή μας. Και με την έκθεση αυτή Έχουμε ένα πολύ καλύτερο εργαλείο για να ε, παρακολουθήσουμε τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας ε, και να σας δώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Θα ήθελα να ε, τονίσω γιατί για, την, για τον οργανισμό θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων είναι τόσο σημαντικό το θέμα των Ρωμά. Όχι επειδή η Κομισιόν ή το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο μας ζήτησαν να υποβάλουμε στοιχεία, αλλά όπως ε, τονίζει και η σύσταση ε, της Κομισιόν, η ένταξη των Ρωμά αποτελούν πρόκληση για το πρόγραμμα Ευρώπη 2020. Η ένταξη των Ρωμά δεν είναι θέμα μειονότητας με την παραδοσιακή έννοια. Εάν κοιτάξουμε τα δικαιώματα των μειονοτήτων που θεσπίζονται σε συνθήκες ή σε συντάγματα. Ε, βλέπουμε ότι διαφέρει το θέμα από το θέμα των Ρωμά. Το θέμα των Ρωμά είναι μια κρίσιμη δοκιμή για την Ευρώπη να αποδείξει ότι μπορεί να ε, αντιμετωπίσει το θέμα της κοινωνικής ένταξης στο σύνολό της. 20 ε, εκατομμύρια άνθρωποι πρέπει να ξεφύγουν από την φτώχεια και τον αποκλεισμό μέχρι το 2020 και η κοινωνική ένταξη των Ρωμά, της, η, μεγαλύτερη ε, εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, είναι απαραίτητη αν θέλουμε να πετύχουμε τους τρεις βασικούς μας στόχους, να έχουμε ευφύ, βιώσιμη ε, και ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το θέμα της φιλετικής διάστασης, διότι αλλιώς επηρεάζονται οι άντρες και αλλιώς οι γυναίκες των Ρωμά. Και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό για να αναπτύξουμε τις πολιτικές ε, που θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές. Η πρόκληση της ένταξης των Ρωμά γενικά ήδη από το 2000 περίπου και μετά όταν οι διεθνείς οργανώσεις άρχισαν να εξετάζουν πιο αναλυτικά το θέμα αυτό και άρχισαν να ξεφεύγουν από τη ρητορική και να βλέπουν τι μπορεί να γίνει πρακτικά. Η πρόκληση λοιπόν είναι ότι η απομόνωση των Ρωμά, ο αποκλεισμό του ε, είναι ένα πρόβλημα με πολλές διαστάσεις, ε, είναι συνδυασμός διαφόρων προβλημάτων ε, και ουσιαστικά εδώ επικαλύπτονται δύο τομείς, η φτώχεια και το θέμα των, δικαιωμάτων, των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν η δουλειά μας εξετάζει και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και το πώς μπορούν να βελτιωθούν αυτές και ταυτόχρονα εξετάζουμε και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι οι διακρίσεις, ο ρατσισμός, η συνειδητοποίηση των ε, ε, δικαιωμάτων ε, και η συμμετοχή στην κοινωνία. Όσον αφορά τα δεδομένα, τα δεδομένα που θέλω να σας παρουσιάσω σύντομα προέρχονται από την μελέτη για τους ΣΕΡΟΜΑ που πραγματοποιήθηκε το 2011 η ειδική ομάδα στην οποία συμμετείχε ο Οργανισμός Θεμελιωτών Δικαιωμάτων. Ήταν μια ομάδα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τον Δεκέμβριο του 2012 ανέφερε ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων και γι' αυτό ε, σχεδιάσαμε μια μελέτη η οποία θα καλύπτει κράτη-μέλη και στην Ανατολή και στη Δύση της Ευρώπης. Είχαμε μελέτες του, της UNDP και από άλλους οργανισμούς. Αλλά δεν, υπήρχαν μέχρι, δεν υπήρχε μέχρι τότε μία μελέτη που να καλύπτει και τις ανατολικές και τις δυτικές χώρες. Και που να δει ποιες είναι οι διαφορές. 11.000 ε, σχεδόν Ρώμα και 5.500 ε, μη Ρώμα επελέγησαν ε, τυχαία και Θέλαμε να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες ε, για να δούμε μήπως οι μη Ρωμά διαφέρουν σημαντικά ε, σε, όσον αφορά τις κοινωνικο-οικονομικές τους συνθήκες αλλά και με τον ε, τρόπο που απολάβουν δικαιωμάτων ή αντιμετωπίζουν θέματα διακρίσεων κοιτάξαμε λοιπόν ε, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και την στέγαση, αλλά θέλαμε να κοιτάξουμε και τα χαρακτηριστικά των οικοκυριών, ε, των γειτονιών ε, και να εξετάσουμε και θέματα ενεργού συμμετοχής στην πολιτική ζωή κλπ συντοποίηση των δικαιωμάτων. Ζητήσαμε από το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής να μας υποβάλουν εκθέσεις από τα 28 κράτη-μέλη με βάση δευτερεύοντα στοιχεία. Με βάση δηλαδή ε, τι, τα, τις υπάρχουσες έρευνες, ε, τις έρευνες που ήδη είχαν γίνει. Ε, από... Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στις κάτω χώρες, τους ταξιδιώτες, τι γίνεται στο Βέλγιο. Τα θέματα αυτά αναφέρονται στις εκθέσεις αυτές και είναι θέματα τα οποία έχουμε θίξει στο παρελθόν και που συμπεριλαμβάνονται και στους στόχους μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι σημαντικό με αυτήν την έρευνα είναι ότι δεν είναι έρευνα όπου ρωτάμε ανθρώπους που επιλέγησαν από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δεν ρωτάμε ανθρώπους που συναντήσαμε στο δρόμο. Έχουμε κάνει μια επιστημονική τυχαία επιλογή ε, που καλύπτει το σύνολο της χώρας. Ε, να σας δώσω παραδείγματα από κάποιες χώρες, από την Τσεχία. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να το δείτε εδώ πέρα, αλλά βλέπετε κάποιες πράσινες κουκίδες, οι οποίες είναι οι τόποι, οι δήμοι όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Οι μαύρες κουκίδες είναι άλλες κοινότητες όπου ζουν οι Ρωμά, οι οποίες όμως δεν επιλέγησαν. Αυτές που επιλέγησαν τυχαία είναι οι πράσινες. Εντός κάθε κοινότητας, εντός κάθε δήμου, πραγματοποιήθηκε τυχαία επιλογή νοικοκυριών, όπου έγιναν συνεντεύξεις και 45 ε, λεπτά με μία ώρα κράτησε η κάθε συνέντευξη. Να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε χάρτη με τους σχετικούς δήμους ε, στη Γαλλία. Στη Γαλλία εξετάσαμε τους gens de voyage, τους ε, ταξιδιώτες, καλύψαμε με διαφορετική μεθοδολογία όμως και αυτό δεν τους έχουμε συμπεριλάβει σε αυτά τα αποτελέσματα, Ρουμάνους μετανάστες καταγωγής Ρωμά. Εδώ λοιπόν ε, βλέπετε ε, τους ε, τόπους όπου διαμένουν αυτοί οι ταξιδιώτες. Η Ισπανία. Όπως βλέπετε και εδώ προσπαθήσαμε να καλύψουμε το σύνολο της χώρας, τα καταφέραμε, δεν είχαμε λοιπόν το σύνηθες ε, δείγμα του Νότου. Έχουμε καλύψει και άλλες ε, περιοχές της Ισπανίας. Προχωράμε στα αποτελέσματα. Να ξεκινήσω από την εκπαίδευση και μάλιστα χωρίς ε, να προχωρήσω κατευθείαν σε ανάλυση αναφύλο. Όσον αφορά τον αναλφαβητισμό, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν να γράφουν και να διαβάζουν. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση σε 8 από τα 10 κράτη-μέλη που ε, εξετάσαμε. Ε, στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 αυτή είναι πολύ σοβαρή ε, κατάσταση, διότι σημαίνει ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες απασχόλησης των ανθρώπων αυτών. Μπορεί όμως να είναι και ένας παραγόντας που συμβάλλει σε σοβαρές μορφές εκμετάλλευσης στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, εκμετάλλευση από ε, κλιματικές οργανώσεις, ε, καταναγκασμός ε, να τους καταναγκάζουν να ζητιανεύουν, εμπορία ανθρώπων, πορνεία κλπ. Αυτή λοιπόν η έλλειψη εκπαίδευσης είναι παράγοντας που εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε, ακ... σε ακραίες περιπτώσεις στόχιας, ακραίες συνθήκες στόχιας. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τους ε, άντρες και τις γυναίκες όσον αφορά τον αναλφαβητισμό, βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε κάποιες χώρες όμως ε, και όχι στο σύνολο των κρατών μελών. Εάν κοιτάξουμε το σύνολο των χωρών, ε, η διαφορά είναι περίπου 10%. Οι γυναίκες Ρωμά έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από ότι οι άντρες. Αν κοιτάξετε όμως την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, οι ε, διαφορές είναι πολύ μεγαλύτερες. Τα καλά νέα είναι ότι αν αναλύσουμε τα στοιχεία αυτά και θα ήταν πολύ πολύπλοκο να σας το παρουσιάσω εδώ, μπορείτε να το διαβάσετε όμως στην ανάλυση που έχω διανύμει, ε, αν εξετάσουμε τις διάφορες ηλικιακές ομάδες θα διαπιστώσουμε ότι ε, οι νέοι βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αυτό λοιπόν αποτελεί καλό νέο. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες ε, λοιπόν ε, η κατάσταση βελτιώνεται και αποφασίσαμε να εξετάσουμε τις γυναίκες Ρωμά ηλικίας 16 έως 24 ετών και βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο έχουν φτάσει το ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης με τους άντρες. Ε, η μεγαλύτερη αύξηση στις διάφορες ηλικιακές δοχμάτες ε, εμφανίζεται στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Ωστόσο σε μία χώρα, την Ελλάδα, παραμένει κρίσιμη η κατάσταση και μόνο το 65% των γυναικών και ανδρών Ρωμά ηλικίας 16 έως 24 ε, μπορούν, ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν οι περισσότεροι. Σημαντική μειοψηφία λοιπόν ακόμα συνεχίζει να μην γνωρίζει και ανάγνωση. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, εδώ βλέπουμε αυτούς που ε, έχουν πάει σχολείο και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να δείτε τα συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά από αυτούς ε, που πήγαν σχολείο τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μεγάλο ποσοστό πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου, το οποίο το βλέπετε εδώ με σκούρο μπλε. Με σκούρο μπλε βλέπετε αυτούς που σταμάτησαν πριν τα 16. Και μιλάμε για τη νέα γενιά ανθρώπους ηλικία 16 έως 24. Αυτή λοιπόν είναι η γενιά που τώρα μπαίνει στην αγορά εργασίας. Ε, για κάποιες χώρες βλέπετε το κίτρινο που δείχνει αυτούς που ποτέ δεν πήγανε σχολείο και είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τις διαφορές σε κάποιες ανατολικές χώρες όπως είναι η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, αλλά και στην Ισπανία βλέπουμε ότι ο αριθμός αυτών που ποτέ δεν πήγαν σχολείο είναι σχεδόν μηδενικός. Έχουν πάει σχολείο λοιπόν, εάν δούμε όμως την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Γαλλία ή την Πορτογαλία, βλέπουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που εγκατέλειψαν το σύστημα και δεν πήγαν σχολείο. Σημαντικό όμως ε, σημαντικό είναι και το μπλε ποσοστό, διότι είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο και μπορεί να μην μπορέσουν να αποσχοληθούν. Υπάρχουν και εδώ σημαντικές ε, διαφορές αναχώρα, αλλά ε, γενικά Περισσότερες ε, γυναίκε Ρωμά εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ηλικία των 16 από ότι άντρες και λιγότερε συνεχίζουν τη διεκπαίδευση μετά τα 16. Η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα με την ε, απασχόληση και τις δυνατότητες ε, απασχόλησης. Εάν δούμε λοιπόν την απασχόληση των γυναικών Ρωμά, βλέπουμε ότι εδώ αντικατοπτρίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης ε, αλλά και των διακρίσεων. Για τις γυναίκες ε, δηλαδή αντικατοπτρίζεται ε, η μη ύπαρξη φροντίδας για τα παιδιά, για παράδειγμα. Βλέπουμε όμως ότι τα μοτίβα αυτά διαφέρουν αρκετά από αυτά που ισχύουν για, το, την πλειοψηφία του πληθυσμού. Ε, γενικά, ε, σημαντικό ποσοστό Ε, το 25% των γυναικών ε, εργάζονται, ενώ το 25% εργάζονται. Ε, το 24% των γυναικών φροντίζουν το σπίτι, ενώ 1% των ανδρών. Σημαντικό όμως είναι εδώ να δούμε ότι σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης οι γυναίκες Ρώμα ε, συμμετέχουν ε, ίσα ή ακόμα και περισσότερο από τους ε, άνδρες όσον αφορά την πληρωμένη εργασία, την αμοιβόμενη εργασία. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί πιθανότατα από το κόστος ευκαιρίας όπως το ονομάζουμε. Μία γυναίκα Ρωμά που θα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι, που θα πρέπει να αφήσει τα παιδιά σε κάποιον άλλο, θα το κάνει μόνο εάν το είδος εργασίας που μπορεί να βρει είναι καλύτερο, εάν δηλαδή είναι πλήρης η απασχόληση. Ε, στο ε, σχεδιάγραμμα αυτό λοιπόν βλέπετε τις γυναίκες και τους άντρες Ρωμά που ε, έχουν αμοιβόμενη εργασία. Σε σκούρο μπλε βλέπετε αυτούς που έχουν πλήρη απασχόληση, σε μεγαλάζιο αυτούς που έχουν μερική απασχόληση, με κίτρινο αυτούς που έχουν δουλειές ad hoc, περιστασιακές και με πράσινο του αυτοαπασχολούμενου. Ε, και είναι σημαντικό εδώ να γνωρίζουμε τι διαφορέ, και αυτό τονίζει ακριβώς ε, το διαφορετικό καθεστώ και τα διαφορετικά θέματα που αντιμετωπίζουν ε, οι κοινότητε Ρωμά σε διάφορε χώρε. Σε χώρες, για παράδειγμα, όπω είναι η Ρουμανία, η Ελλάδα ή η Βουλγαρία, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανδρών αλλά και γυναικών που εργάζονται σε περιστασιακές δουλειές, ενώ πολύ χαμηλό ποσοστό ανδρών και γυναικών εργάζονται σε ε, θέσεις πλήρους απασχόλησης, αλλά αυτό αλλάζει αν κοιτάξουμε τις ε, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ε, το μεγάλο κενό υπάρχει στις υπαίθριες περιοχές και το μεγαλύτερο κενό, η μεγαλύτερη διαφορά υπάρχει σε ανθρώπους που ζουν σε καταβλισμούς, ιδιαίτερα στην Ιταλία. Η επόμενη διαφάνεια. Ενδιαφέρουσα είναι η σχέση ανάμεσα ε, στην ε, δραστηριότητα και στην οικογένεια. Όταν ε, ρωτήσαμε τους όταν ρωτήσαμε σχετικά με τα μέλη του νοικοκυριού, ρωτήσαμε άσχετα από την ηλικία εάν ζουν σε κάποιο είδους γάμου παραδοσιακού, νόμιμου ή συγκατοίκηση το 2% όσων απάντησαν, το 2% των παιδιών ε, στον οικοκυριό πράγματι σε ηλικίας 10 έως 15 ετών ε, ήταν παντρεμένα με κάποιο τρόπο, πολύ χαμηλό ποσοστό, ωστόσο υπήρχαν. Εάν κοιτάξουμε τα κορίτσια των Ρωμά ηλικίας 16 με 17, βλέπουμε πιο ε, ψηλά ποσοστά. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε το θέμα της εκπαίδευσης. Οι γυναίκες που που ήταν ε, παντρεμένες ε, ή συγκατοικούσαν όταν ε, σε σύγκριση με όλα τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας είχαν λιγότερο την τάση να παραμένουν εντός του εκπαιδευτικού συστήματα, συστήματος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχει συνέπειες στις, ευκαιρίες, στις μελλοντικές τους ευκαιρίες. Η επόμενη διαφάνεια. Όσον αφορά την υγεία, και αυτό αναφέρθηκε νωρίτερα, βλέπουμε να υπάρχει διαφορά, όχι ανάμεσα στις γυναίκες και τους άντρες των Ρωμά. Ε, εδώ περισσότερο οι άντρες Ρωμά λένε ότι είναι ε, κακή η κατάσταση της υγείας τους. Εάν συγκρίνουμε όμως τις ε, γυναίκες των Ρωμά με τις γυναίκες μη Ρωμά, βλέπουμε σημαντική διαφορά όσον αφορά αυτές που λένε ότι η κατάστασή, τους, ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι κακή ή πολύ κακή. Όταν εξετάσαμε την ε, φαρμακευτική ασφάλιση, ρωτήσαμε αν γνωρίζουν αν έχουν φαρμακευτική ασφάλιση. Βλέπουμε λοιπόν ε, σημαντική διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες Ρωμά και τις ε, άλλες γυναίκες. Ακόμα και αν είναι ασφαλισμένες δηλαδή, το να μην γνωρίζουν ότι είναι ασφαλισμένες μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους, ε, διότι σημαίνει ότι δεν θα, δεν θα πηγαίνουν στο γιατρό ε, να πάρουν συμβουλές ε, και δεν θα προσέχουν την υγεία τους. Θα πρέπει να περάσουμε πολύ γρήγορα μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια που δείχνει τις στεγαστικές συνθήκες και Έχουμε χρησιμοποιήσει τα τρία βασικά κριτήρια, ε, ηλεκτρισμό, αποχέτευση και ε, τρέχον είδωρ. Ε, αυτά συνδέονται άμεσα με θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, καθώς και το κόστος της στέγασης. Εάν συγκρίνουμε όμως νοικοκυριά Ρωμά και μη Ρωμά, οι διαφορές, όπως είπαμε στο παρελθόν, είναι πολύ σημαντικές μεγάλες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά πιο συχνά ζουν σε πολύ κακές συνθήκες στέγασης. Και να κλείσω με την τελευταία διαφάνεια για την φτώχεια. Εδώ έχω προσθέσει και τα αποτελέσματα για τον Εθνικό Μεσόρο της Eurostat. Βλέπουμε ποιοι κινδυνεύουν να ζουν υπό συνθήκες στόχιας δηλαδή που ζουν ε, σε νοικοκυριό με εισόδημα ε, χαμηλότερο του 60% ε, του εθνικού μέσου όρου. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν πολλά να γίνουν για να ε, έχουμε ισότητα και οι διαφορές ανάμεσα στους ε, Ρωμά και τους μη Ρωμά που μένουν ε, σε γειτονικέ περιοχές, αλλά και σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό που βλέπετε εδώ με κόκκινο, δείχνει ότι απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να πετύχουμε να, ε, ε να σώσουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια μέχρι το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, επειδή τελειώνει ο χρόνος θα ήθελα να ζητήσω 5 λεπτά υπομονής από τους διερμηνείς. Έτσι ώστε να μπορέσει η Κίνγκα Γκόντς να κάνει τα τελευταία της ε, σχόλια και να ολοκληρώσουμε. Πέντε λεπτά. Ναι, λυπάμαι πολύ που δεν έχουμε χρόνο. Αυτό συμβαίνει συχνά. Έχουμε πολλές πληροφορίες και λίγο χρόνο. Είμαι σίγουρη πως ε, αυτή η έρευνα που είδαμε, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα Εάν θέλουμε ισχυρέ δεσμεύσει από τα κράτη-μέλη, πρέπει να δούμε και αυτέ ε, τι διαφάνειε και αυτά τα στατιστικά στοιχεία, να δούμε τι γίνεται με την εκπαίδευση, με τη στέγαση και ελπίζω η κατάσταση αυτή να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Η παρουσίαση αυτή όμως ε, και γενικά η σημερινή συνεδρίαση κατέστησε σαφέ ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχει γίνει κάποια πρόοδο σε ορισμένου τομεί, στην απασχόληση για παράδειγμα, στην εκπαίδευση. Αυτό που χρειάζεται όμω είναι να καταλάβουν όλοι ότι η ένταξη των Ρωμά δεν είναι μόνο κάτι που αφορά του Ρωμά και μόνο, είναι κάτι που αφορά όλου. Εάν συνεχίσουν οι διακρίσει και οι προκαταλήψει, τότε δεν θα αρκέσει να έχουμε περισσότερους ε, μορφωμένους νέους ε, Ρωμά διότι δεν θα μπορούν μετά να βρουν δουλειά. Πιστεύω λοιπόν πως ε, τουλάχιστον για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ημέρα. Πιστεύω να ήταν και για σας, ελπίζω να ήταν και για σας και ελπίζω να έχουμε σωστές και ισχυρές συστάσεις που θα προκύψουν από όλη την ε, συνεισφορά όλων των ε, συμμετεχόντων. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Όποιος θέλει, να σχολιάσει. Παρακαλώ. Ναι, βρήκα τις στατιστικές αυτές αρκετά ενδιαφέρουσες και αν κατάλαβα καλά, κάποιες από αυτές ήταν και κάτι που προκάλεσε έκπληξη κιόλα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία ανάμεσα στην ε, Ανατολική ε, ευρώ όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση στην Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό θα, που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν έχετε κάποιο... Κάποια πρώτον, κάποια αντίγραφα όλων αυτών και δεύτερον κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Διότι θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να τα κοιτάξω με την ησυχία μου. Μας ε, δώσατε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και η σύνοψη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά θα ήθελα να ξαναδώ τις ε, διαφάνειες αυτές. Ναι, καταρχάς έχουμε υλικό και υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και είναι στη διάθεσή σας. Και εκεί ενδεχομένω να βρείτε και ορισμένες εξηγήσει για το γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Εμείς αυτό που θέλαμε να δείξουμε είναι να κάνουμε μια απεικόνιση της κατάσταση, να γίνει μια ποιοτική ει βάθο έρευνα που με αφορμή αυτή να καταλάβουμε γιατί ε, έχουν συμβεί αυτά. Αυτό που ζητάτε εσείς είναι κάτι που θα εμβαθύνει πολύ περισσότερο και αυτό δεν γίνεται με αυτήν την ε, μελέτη που έχουμε εκπονήσει εμείς. Χρειάζεται μια άλλη ε, μελέτη η οποία θα αρχίσει από του χρόνου και θα συμπεριλάβει πολλές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις αιτίε και τα αποτελέσματα. Υπάρχουν άλλα σχόλια, άλλες μαρτυρίες, άλλες ερωτήσεις. Έχετε ήδη λάβει το λόγο μία φορά. Δεν θέλω να το κάνω αυτό στους διερμηνείς, να σας ξαναδώσω το λόγο. Παρακαλώ, κάποιος άλλος. Ναι, οι διερμηνείς κανονικά δουλεύουν μέχρι τις 6 και μισή, αλλά έχετε δίκιο. Ας το κάνουμε. Ναι, νομίζω πως ε, στις κάτω το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ότι ε, οι άνθρωποι αυτοί δεν, ε, γίνονται, δεν γίνονται δεκτοί ούτε ως Ρωμά, ούτε ως Σύντη, ούτε ως τάξη διώτες. Δεν γίνονται αποδεκτοί λόγω της κουλτούρας τους, λόγω του τρόπου ζωής τους. Και επίσης θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ελέγχους για το αν τα κονδύλια που διατίθεται για τους ε, Ρωμά πραγματικά φτάνουν μέχρι εκεί. Διότι πολλές φορές ε, και μάλιστα σχεδόν πάντα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ελέγξετε εάν τα κονδύλια που διατίθεται για βοήθεια μας βοηθάνε πραγματικά. Ναι, δεν θα υπήρχε καλύτερο κλείσιμο για όλη αυτή την ε, η Μερίδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε σε επαφή μαζί μας και οι βευροβουλευτές που συνεργάζονται για αυτή την έκθεση και οι υπόλοιποι που ενδιαφέρεστε. Οι επόμενες πέντε εβδομάδες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όσοι πάλι ενδιαφέρεστε, έχετε όλα τα έγγραφα στη διάθεσή σας να τα διαβάσετε. Η έκθεση αυτή θα είναι πολύ σημαντική, θα είναι πολύ βαριά. Η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή στην Επιτροπή θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και Ελπίζουμε να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου και αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ζωντανά. Έχουμε λίγες εβδομάδες, σας παρακαλώ λοιπόν να, το, να φροντίσετε να γίνει εκθέσεις πιο δυνατή γίνεται. Ευχαριστώ.